Κύριε Ντουκαζόλιομι, ε, συνειδητοποίησατε ότι σας χειροκρότησαν όταν μπήκατε στην αίθουσα. Γιατί, ξέρετε, γιατί είστε ο μόνος ευρωβουλευτής. Είναι κρίμα, πραγματικά. Τι να πω, ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία. Πάντως, ετοιμαζόμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα τρομακτικά ενδιαφέρον με πολλούς εμπειρογνώμονες εμπειρογνώμονες από τη Ουάσιγκτον μεταξύ άλλων για να μας μιλήσουν για το ρόλο των ιδιωτικών στρατιωτικών ε, εταιριών και των ιδιωτικών εταιριών ε, ασφάλειας. Είναι το πρώτο μας σημείο. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό καταρχήν και συνεχεία θα συζητήσουμε μια μελέτη για την ελευθερία έκφρασης και τη σκεφτική ελευθερία. Θα μα την παρουσιάσουν και εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει μία επιτροπή. Θα κάνει μια ανταλλαγή απόψε με εκπροσώπους μιας της υποομάδας για την οικοδόμηση θεσμών ε, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καμπότζης. ήθελα να συμμετάσχουμε όλοι λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση. Ανακοινώσει τη Προέδρου, σημείο 2. Αν σα ικανοποιεί η μερίσια διάταξη, θα υιοθετήσουμε στι 18 σε 8 Δεκεμβρίου ζητήσαμε ένα ψήφισμα να υιοθετηθεί, υιοθετήσαμε άλλο ένα ψήφισμα για τη Ζιμπάμπουε. Το Συμβούλιο αποφάσισε να διευρύνει τον κατάλογο προσώπων που αφορά το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και για τα οποία μειώνεται ή απαγορεύεται η υποδοχή τους, η εισδοχή τους στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το ζητήσαμε και αυτό με ψήφισμα και σήμερα είναι και Ε, δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Μάθατε για την ε, συνοπτική εκτέλεση του δύο ατόμων, ο ένας ε, δικηγόρος και μια κυρία που είναι δημοσιογράφος, ε, δούλευε στο, στην ίδια εφημερίδα της Άννας Πολιτόσκαβια. Θα συζητήσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία επευκαιρία ενός νέου γύρου διαβουλεύσεων που θα γίνει στις 30 Μαρτίου και θα προετοιμάσουμε αυτή τη συνάντηση στις 2 Μαρτίου στη συνεδρίασή μας. Κάτι άλλο τώρα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την άσχημη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τινησία. Τις τελευταίες εβδομάδες, ε, όπως ε, συμβαίνει συνήθως, μία εκστρατεία συκοφαντίας της κυρίας Σιέμπεζετρής που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα της είναι πολύ γνωστή στην Τινησία. Υπάρχει μία ενόχληση και μία πίεση των δημοσιογράφων του ραδιοφώνου Καλιμά που δεν λειτουργεί πια σήμερα. έχουν κλείσει τα γραφεία, όλοι οι υπολογιστέ και όλο το υλικό του ραδιοφωνικού σταθμού κατασχέθηκε από την αστυνομία είναι μια απαράδεκτη παραβίαση, ακόμα μία, ε, εναντίον της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης στη χώρα αυτή. Στις 23 επίσης ε, Ιανουαρίου, ο κ. Σαμίν που είναι συντονιστής για ανθρώπινα δικαιώματα στο Μαγκρέμπ, είχε ραντεβού ε, με μέλη της την ισιακής κυβέρνησης, αλλά δεν μπόρεσε, το απαγόρευσαν να έρθει σε επαφή. Ζήτησε από τον Πρόεδρο να κάνουμε κάτι, μια πρωτοβουλία για τη χώρα με αντικείμενο τη χώρα αυτή. για να δούμε τι θα γίνει και με τις σχέσεις μας μεσοπρόθεσμα με τη χώρα αυτή. Η χώρα μας ανησυχεί βεβαίως ό,τι αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ ωραία. Δύο μικρόφωνα μου δίνετε. Πάμε στην ανταλλαγή απόψεων στο σημείο 3 για το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ιδιωτικέ στρατιωτικέ εταιρείε και ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση με του εμπειρογνώμονε για του κανόνε που διέπουν τι δραστηριότητε των εταιριών αυτών και τι παραβιάσει έχουν σημειωθεί από τι εταιρείε αυτέ που έχουν διαφορετικές δραστηριότητες, επιμελητιακή βοήθεια, κατάρτιση των εθνικών τακτικών στρατών, παροχή ασφάλειας κτλ. Έχουμε συχνές παραβίασεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερβολική άσκηση βίας κατά των αμάχων, απάνθρωπη μεταχείριση, εξαναγκαστική πορνεία, ε, σεξουαλικά εγκλήματα, εκβιασμός, μη σεβασμός της ε, ουδετερότητας, της ε, κυριαρχίας των ατόμων, δολοφονίες, απίστευτες παραβιάσεις και πολυάριθμες. Παράλληλα, οι κανόνες που διέπουν τις δραστηριότητε τους θα πρέπει να αναδιατυπωθούν σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Έχουμε εδώ τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε τον κύριο Κίνση, τον κύριο Μεσνέρ και τον κύριο Κολανόφσκι. Για να δούμε πώς μπορούμε να ελέγξουμε, θα δούμε τι κανόνες μπορούμε να εφαρμόσουμε σε αυτές τις εταιρείε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κίνση από το King's College ε, στο Λονδίνο του Τμήματος ε, Αμυντικών Σπουδών. Θα μας κάνει μια παρουσίαση 10 λεπτών. Κύριε Κίνση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εστιάσω τις, ε, την παρουσίασή μου κυρίως ε, στις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας και όχι τις ιδιωτικές ε, στρατιωτικές εταιρείες που είναι ένα σώος που χρησιμοποιούν περι, κυρίως οι Αμερικάνοι. Οι περισσότερες εταιρείες δίνουν όχι στρατιωτική υποστήριξη αλλά ασφάλεια. Θέλω να εστιάσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι μπορεί να κάνει και τι κάνει και στις εταιρείε που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι αυτές που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο συνάδελφος θα μιλήσει για τις υπόλοιπες. Ξεκίνησε αυτός ο κλάδος στις αρχές της δεκαετίας του 70 και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παροχή ιδιωτικής ασφάλειας ε, έγινε θέμα και ζήτημα μόνο στη δεκαετία του 1990 ε, με τις επιχειρήσεις στην Αγκόλα και στη Σιέρα Λεόνε. Ε, το Human Rights Watch έγραψε μια έκθεση για το θέμα της παραβίασης των δυνάμεων της Σουνιτά και στην έκθεση αυτή δεν εντοπίστηκαν ε, παραβιάσεις των δικαιωμάτων από εταιρείε, αλλά Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήταν, η δουλειά αυτών των εταιριών ήταν ε, παροχή προστασίας. Τα πράγματα άλλαξαν μετά το δεύτερο, με τον ψυχρό πόλεμο. Οι εταιρείε δίνουν περισσότερες υπηρεσίε, υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ίσως και περισσότερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο Ιράκ προστατεύουν τις αυτοκινητοπομπές, ε, δίνουν φρουρούς, Επειδή εμπλέκονται περισσότερο, υπάρχουν ε, περιθώρια για μεγαλύτερε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για ένα μικρό αριθμό εταιριών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι περίπου 30 ή 40 εταιρείε αυτέ που είναι αρκετά μεγάλε. Είναι εύκολο να δημιουργήσει κανεί μια εταιρεία. Χρειάζεται ένα φαξ και τη δυνατότητα να συνάψεις κυβερνητικές ε, συμβάσεις. Έτσι ξεκινάνε αυτές οι εταιρείε. Μιλάμε λοιπόν για ένα μικρό αριθμό εταιριών για το πώς θα ρυθμίσουμε τις δραστηριότητε τους. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείε ε, δίνουν, εξασφαλίζουν την ε, ασφάλεια χωρίς τη χρήση όπλων. Uh, Οι περισσότερες εταιρείε δουλεύουν εκεί σε, σε χώρες όπως το Κονγκό, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η Σομαλία, όπου δεν μπορούν να λογοδοτήσουν. Σε περισσότερες ε, περιπτώσεις όμως ε, δουλεύουν στην Τανζανία, στην Κένια κτλ. οτιδήποτε πάει στραβά πρέπει να λογοδοτήσουν. Γιατί υπάρχουν κοινωνικά συστήματα σε αυτέ τι χώρε που, πρέπει, που του υποχρεώνουν να το κάνουν. Τώρα, στο Ιράκ δουλεύουν για πρεσβείες, ε, προστατεύουν το προσωπικό των ε, πρεσβειών, για την κυβέρνηση του Ιράκ, για διάφορους φορείς και οργανισμούς του ΟΗΕ, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, Προστατεύουν επίσης ε, στελέχη εταιριών, την KBR, παραδείγματο χάρη. Η Aegis, ε, μια άλλη εταιρεία, ε, βοηθάει στην οικοδόμηση του Ιράκ, προστατεύει αξιωματούχους Αμερικανούς, μηχανικούς, στρατιωτικούς, στελέχη επιχειρήσεων, όλους αυτούς που συνεργάζονται για να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Έχουν μεγάλες, μεγάλα συμβόλαια αυτές οι εταιρείε και συγκεκριμένα οι Aegis. Επίσης ε, καταρτίζουν την, τους Ιρακινούς αστυνομικούς και βοηθάει για να καταρτιστεί ο στρατός του Ιράκ. Η Aegis ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των εκλογών το 2005 που έγινε στο Ιράκ. Τέτοια δουλειά κάνουν στο Ιράκ λοιπόν. Σε άλλα μέρη του κόσμου παρέχουν προστασία και μεταρρυθμίζουν το τομέα της ασφάλειας. Επίσης, υπάρχουν προστασία σε αυτοκινητοπομπές ε, στο Ιράκ κυρίως. Η μελλοντική αγορά τώρα του κλάδου. Ο κλάδος αυτός ε, δεν θα λέω ότι φθήνει, είναι λάθος λέξη αυτή. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο ανώτατο όριο ε, μάλιστα έφτασε τότε το 2006-2007. Από τότε υπάρχει μια πτώση, αν θέλετε, της δουλειάς. Επομένως, τρέφονται αλλού τώρα, σε άλλους τομείς, σε άλλες αγορές. Σταθε, σταθερότητα ε, μετά τους πολέμους, ε, ανθρωπιστικός τομέας, ε, αναπτυξιακός τομέας, είναι οι τομείς που αυτός ο κλάδος θεωρεί ότι μπορεί να ενεργοποιηθεί στο μέλλον. Και εδώ πρέπει να δούμε τι πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να προκύψουν από αυτές τις εταιρείε. Σε μέρη όπως το Ιράκ, είναι δύσκολο να προσμετρήσουμε το επίπεδο των παραβιάσεων. Και στο Αφγανιστάν το ίδιο. Υπάρχουν μερικές ε, γνωστές περιπτώσεις που είναι γνωστές ε, στα και προβλήθηκαν από τα ΜΜΕ, Παραδείγματο χάρη Abu Ghraib. Έχουμε δύο ή τρει περίπου τέτοιε γνωστέ περιπτώσει, αλλά υπάρχουν και άλλε παραβιάσει από τέτοιε εταιρείε στο Ιράκ τα τελευταία πέντε χρόνια. Αλλά σε ποιο βαθμό κανένας δεν ξέρει ακριβώς. Και αυτό είναι μείζον πρόβλημα Ξέρουμε ότι ορισμένε από τι εταιρείε ε, παραβίασαν ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά οι περισσότερε, σε μία από μία τις εκθέσεις που έχουν γραφτεί αναφέρθηκε ότι συμπεριφέρονται σωστά και διατηρούν υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές. Αυτή την έκθεση την ε, δημοσιεύτηκε πέρυσι για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, τι νομικά εργαλεία που μπορούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διώξουμε όσους παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν οι, ο ορισμός ε, για τους μισθοφόρους ή ο νόμος κατά των μισθοφόρων. Στο διεθνό δίκαιο ορισμός του μισθοφόρου, για να το πω ομά, είναι λίγο άχρηστος για να διώξουμε ε, τις ιδιωτικές εταιρείες. Ένα μελετητής είπε ότι ότι ποτέ δεν έχει διωχθεί κάποιος ε, από τις εταιρείε αυτές ε, με αυτόν τον ορισμό. Γιατί μπορούμε να τον παρακάμψουμε πολύ εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια. Ένα άλλο διεθνέ εργαλείο είναι η Διεθνή Σύμβαση κατά τη ε, στρατολόγηση, χρήση, χρηματοδότηση και εκπαίδευση των μισθοφόρων. Του 89. Ε, τέθηκε σε ισχύ το 2001, αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για να διώξουμε τελικά τους μισθοφόρους. Οι μόνο δύο ήταν Σάιμον Μαν και Νίκ Ντετόιτ, που είναι τώρα στη φυλακή στην Γουινέα. Το 2002 η Βρετανική κυβέρνηση υιοθέτησε την πράσινη βίβλο για να απαντήσει σε μια υπόθεση την υπόθεση Sandlight του 97-98, που είναι μια ιδιωτική βρετανική εταιρεία που παραβίασε το εμπάργκο όπλων στη Σιέρα Λιόνε. Ε, σε αυτή την πράσινη βίβλο υπάρχουν διάφορες συστάσεις για να ρυθμίσουμε τις δραστηριότητες αυτές. Όμως καμία από αυτές τις συστάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Αυτό το μήνα το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί τελικά να κάνει μια ανακοίνωση για το ποια επιλογή προτιμάει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα. Το άλλο έγγραφο, το οποίο δεν είναι ε, νομικά δεσμευτικό, είναι μια πρωτοβουλία της ελβετικής ε, κυβέρνησης. Και πιο μάλλον πιο συγκεκριμένα του Ερυθρού Σταυρού. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό για τα κράτη, αλλά μιλάει για καλές πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιεί ο κλάδος. Είναι μια καλή βάση για να προχωρήσουμε. Τα κριτήρια, ας πούμε, είναι οι διαδικασίες που να υπάρχουν για να επιλέγουμε ε, τα συμβόλαια, οι όροι των συμβολέων, με αυτές τις εταιρείες κτλ. Είναι θαυμάσιο έγγραφο για να προχωρήσουμε. Θα προχωρήσω γρήγορα επειδή έχω μόνο 10 λεπτά. Η βιομηχανία αυτή υπάρχει, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, να είστε σίγουροι. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε αυτά που συνέβησαν ας πούμε στο Ιράκ μεταξύ του 2004 και 2007. Ένα τεράστιο αριθμό από τέτοιες εταιρείες ε, για να βοηθήσουν στην ε, ανοικοδόμηση. Συχνά ε, παραβίαζαν διάφορους νόμους και ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά ήταν στο απειρόβλητο. Δεν τιμωρήθηκαν γι' αυτά. Η αγορά για τις υπηρεσίες τους είναι παγκόσμια. Αλλά οι δύο βασικές χώρες που εστιάζονται αυτές οι εταιρείες είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Η πρώτη εταιρεία ήταν η WatchGuard International που δημιουργήθηκε από, ένα πρώην, από ένα πρώην μέλος των ε, ειδικών δυνάμεων SAS ε, και είχε έδρα στο Λονδίνο. Τώρα υπάρχουν και σε άλλες χώρες, στη Γαλλία, στο Ισραήλ, στην Αυστραλία και στην Νότια Αφρική, για να φέρω τέσσερις ακόμα. Με βάση την έρευνα που έχω κάνει, βρήκα ότι το να εγκατασταθούν σε αυτές τις χώρες είναι πιο δύσκολο, γι' αυτό ο αριθμός τους είναι πιο μικρός. Στην, στην Ολλανδία, ας πούμε, ε, υπάρχουν δύο τέτοιε εταιρείε, αλλά εγκαθίστανται και σε άλλε εταιρείε, αλλά στο βαθμό που εγκαθίστανται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Η έκθεση του Human Rights Watch λέει, ε, υποδηλώνει ότι οι περισσότερες από αυτές τι εταιρείε σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένω, το θέμα είναι το πώ θα αντιμετωπίσουμε το μικρό αριθμό εταιριών που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει ένας τέτοιος μικρός αριθμός και μικρό αριθμό ανθρώπων που αγνοούν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Από την έρευνα που έκανα, ε, πιστεύω ότι οι κανονισμοί είναι σημαντικοί. Πρέπει να υπάρξουν τέτοιοι κανονισμοί και πρέπει να αφορούν τις δραστηριότητες που είναι η παροχή ασφάλειας μέσω όπλων. Πολλές από τις εταιρείες που θεωρούνται ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας στην πραγματικότητα δίνουν ε, απλώς επιμελητιακή υποστήριξη. Στην πραγματικότητα δηλαδή ε, υπάρχει ένας μετασχηματισμός ε, με τον, για τον τρόπο, με τον τρόπο που λειτουργούν οι στρατοί. Ε, πηγαίνουν δηλαδή από στρατιωτικές δραστηριότητες σε πιο εμπορικές Αυτό είναι τελείως διαφορετικό θέμα από την παροχή ασφάλειας με όπλα. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θελήσει να ρυθμίσει τη δραστηριότητα της KBR, ε, θα έρθει σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ, ας πούμε, που βασίζεται στην, στην επιμελητιακή υποστήριξη της KBR για τις επιχειρήσεις του στο Αφγανιστάν. Η MOD, το Υπουργείο Άμυνας, θα ασχοληθεί με, το... τον, με τον νόμο για τις ανοπλές δυνάμεις. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποιεί τέτοιε ιδιωτικέ εταιρείες, ενώ το Υπουργείο Άμυνα όχι. Νομίζω το ίδιο και το Γαλλικό Υπουργείο Άμυνα. Μόνο τα Υπουργεία Εξωτερικών τα χρησιμοποιούν. Γιατί οι στρατιωτικοί δεν μπορούν να προστατεύσουν τους αξιωματούχους τους. Αυτά, Πρόεδρε. Ελπίζω να μην ξεπέρασα το δεκάλεπτο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κίνση. Τώρα το λόγο δίνουμε στον κύριο Μέσνερ, ο διευθυντής ε, του τμήματος Peace Operations. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την πρόσκληση που μας απέθυνε να μιλήσουμε. Η Ένωσή μα είναι μια οργάνωση που εκπροσωπεί 50 εταιρείε του ιδιωτικού τομέα παγκοσμίω που προμηθεύουν υπηρεσίες ειρήνευση και σταθερότητας. Οπότε ελπίζουμε να μπορέσουμε να σας δώσουμε και τη δική μας σκοπιά. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως όλοι μας εδώ πέρα ω ανθρωπιστέ έχουμε ένα κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε δηλαδή τη λειτουργία των επιχειρήσεων ειρήνης και σταθερότητας για να διαχωρίζονται οι εμπόλεμες πλευρές, να προστατεύουμε τους αμάχους και να υπάρχει σταθερή ειρήνη. Κοινό συμφέρον στο να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα επιτρέψουν σε κοινωνίες ρημαγμένες από τον πόλεμο να ανοικοδομηθούν. Επίσης νομίζω ότι μπορώ να πω πως όλοι μας εδώ πέρα, ως ένα βαθμό, απελπιζόμαστε όταν βλέπουμε επιχειρήσεις ειρήνης και σταθερότητας σε διάφορες χώρες να αποτυγχάνουν. Η πραγματικότητα δυστυχώς τέτοιων επιχειρήσεων σήμερα είναι πως ε, δεν έχουν αρκετή χρηματοδότηση και πόρους. Καθώς οι επιχειρήσεις ε, και του ΟΗΕ και άλλων οργανισμών επεκτείνονται συνεχώς. Οι συνεισφορές των δυτικών κρατών μελών συνεχώς μειώνονται. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ειρήνης και σταθερότητας βασίζονται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και με κάθε σεβασμό σε αυτές τις χώρες η πραγματικότητα είναι πως δεν έχουν την ίδια καλή εκπαίδευση, πόρους και εξοπλισμό όπως οι ε, δυτικοί στρατοί. Υπάρχουν κενά στον επαγγελματισμό και στις δυνατότητές τους και είναι ένα κενό το οποίο πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας και είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τι εννοούμε ακριβώς ιδιωτικό τομέα. καθώς οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ειρήνης και σταθερότητας συμπεριλαμβάνουν αερομεταφορές, βασικές ε, ε υποστηρίξεις, ε, επιμελητεία, μεταφορές, ε, τον ιατρικό κλάδο και βέβαια την ασφάλεια. Οι εκτιμήσεις ε, των ατόμων που απασχολούνται αυτή τη στιγμή στο Ιράκ είναι γύρω στα 160.000 άτομα. Στους 168.000 μόνο 10.000 έχουν ε, ως απασχόληση την ασφάλεια. Να το επαναλάβω. Από το προσωπικό του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζει τις συμμαχικές δυνάμεις στο Ιράκ, λιγότερο από το 10% είναι στον τομέα της ασφάλειας. Όταν μιλάμε για την ιδιωτική ασφάλεια, πρέπει να το δούμε ως ένα μικρό συστατικό κομμάτι ενός πολύ ευρύτερου κλάδου. 160.000 άτομα επίσης ακούγονται πάρα πολλά για ιδιώτες που αλωνίζουν στο Ιράκ, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε κατά νου την ταυτότητά τους και το τι κάνουν. Κάποιοι είναι δυτικοί και κάποιοι είναι από τρίτες χώρες, πάνω από το 80% όμως είναι Ιρακινοί που απασχολούνται στην ανοικοδόμηση της ίδιας τους της χώρας. Το μοντέλο αυτό της εκτενούς απασχόλησης του ντόπιου πληθυσμού νομίζω αντικατοπτρίζεται και επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέρα από τα προφανή ωφέλη, επίσης διασφαλίζει πως ο ντόπι αυτός ένα συμφέρον στην ανοικοδόμηση, δίνει δουλειές και παρέχει και δεξιότητες και βεβαίως δίνονται και σημαντικά οικονομικά ωφέλη για το μέλλον. Εξίσου σημαντικό είναι βεβαίως να έχουμε κατά νου και το οικονομικό μέγεθος του κλάδου. Βεβαίως κάποιες υπερβολικές εκτιμήσεις μιλάνε για 100 δισεκατομμύρια δολάρια είπα, στην πραγματικότητα είμαστε πιο κοντά στο 1 πέμπτο αυτού του ποσού. Επίσης το ποσοστό κέρδους στις περισσότερες συμβάσεις είναι από το 1 έως 3% και μια εταιρεία είναι πολύ τυχερή εάν έχει ένα ποσοστό κέρδους 5%. Δεν είναι λοιπόν ο κλάδος με το μεγάλο κέρδος που ορισμένοι θεωρούν. Πράγματι γίνεται πολλής λόγος για τον ε, κλάδο αυτό. Βεβαίως το εάν αξίζει 100 δισεκατομμύρια ευρώ ή 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με συγχωρείτε αυτός ο κλάδος, εξίσου ε, σημαντική είναι η 20 δισεκατομμυρια δολαρια με συγχωρειτε αυτος ο κλαδος εξισου σημαντικη ειναι η λογοδοσια και η υπευθυνότητα. Η πείρα μας έχει δείξει πως ε, η φύση αυτών των ε, περιβαλλόντων, των συγκρούσεων δηλαδή, συχνά είναι πιο ευεπίφορη στις ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό όμως δεν περιορίζεται σε μία μόνο πλευρά. Οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γίνονται και από τους ειρηνευτές και από τους ε, αντιμαχωμένου και από τον ιδιωτικό τομέα και όταν προσπαθούμε να σταματήσουμε τις μελλοντικέ παραβιάσεις δεν πρέπει να υποθέτουμε πως μόνο μία πλευρά έχει μεγαλύτερη τάση για τέτοιες παραβιάσεις ή χρειάζεται περισσότερη ρύθμιση. Πιστεύω πως όλες οι κατηγορίες δρόντων πρέπει να πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές. Υπάρχουν αρκετοί νόμοι που ρυθμίζουν τα του κλάδου. Οι δε συμβασιούχοι του ΟΗΕ που αναλαμβάνουν επίγοντα συμβόλαια έχουν πάρα πολλού όρου να εκπληρώσουν από τα πολύ απλά πράγματα όπως το να δίνουν αναφορά μέχρι το εμπόριο όπλων και ανθρώπων οι δε πράξεις των μεμονωμένων αυτών συμβασιούχων υπάγονται σε έναν αμερικανικό νόμο στρατιωτικής εξοδεδαφικότητας που προσπαθεί να περιορίσει τις εγκληματικές ενέργειες από αυτούς. Βεβαίως, διεθνώς τα πράγματα δεν είναι τόσο εύρωστα από πλευράς νομοθεσίας, αλλά αυτό δεν είναι ζήτημα των ιδίων των εταιριών, είναι ζήτημα δυναμίας δράσης των διεθνών οργανισμών. Παρ' όλα αυτά αυτό το κενό κλείνει χάρη σε διάφορες εξελίξεις όπως το έγγραφο του Μοντρέ και μια πρωτοβουλία της Ελβετικής Κυβέρνησης και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Πέρα από όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο συχνά ξεχνάμε είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων αυτών και των εταιριών καλύπτονται από τους τοπικούς νόμους. Εκεί όπου χρειάζεται διεθνής νομοθεσία είναι μάλλον οι εξαιρεσει και στις περιπτώσεις αυτές ούτως ή άλλως οι υπήκοοι της ίδιας χώρας που φιλοξενεί και που είναι ο κύριος όγκος των εργαζομένων καλύπτονται από την εσωτερική του νομοθεσία. Π.χ. στο Αφγανιστάν μιλάμε για 99% των εργαζομένων. Όταν μιλάμε για την ασφάλεια βεβαίως η αναζήτηση τελειότητας δεν τελειώνει με τη ρύθμιση. Η επαρκής εκπαίδευση, ο έλεγχος των εργαζομένων και πρακτικοί κανόνες καθώς και εγχειρίδια εκστρατείας είναι εξίσου σημαντικά. Το εάν υπάρχουν ε, αν και υπάρχουν κανόνες βεβαίως στα χαρτιά, πρέπει να εφαρμόζονται. Έχουν υπάρξει κάποια περιστατικά ατυχής, ε, ατυχούς συμπεριφοράς, με συγχωρείτε, στο Ιράκ, καθώς ε, και δράσεις με ατιμορρησία. Δεν πρέπει όμως να μπερδεύουμε την ατιμορρησία με το, τη δυνατότητα επίβλεψης. Συγκεκριμένα στο Ιράκ, έχουμε άτομα τα οποία απασχολούνται για πάρα πολύ μικρό χρόνο και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων. Η στρατιωτική δικαιοσύνη, σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία, κατά κανόνα λειτουργεί, αλλά βεβαίως δεν υπάρχει η σωστή επιβολή. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ε, οι ιδιωτικές αυτές εταιρείες δεν διαφέρουν από τις ιδιωτικές εταιρείες που λειτουργούν σε πιο καθημερινές ας πούμε, καταστάσεις όπως οι δημόσιες μεταφορές ή η τεχνολογία. Τα συμβόλαια πρέπει να επιβλέπονται σωστά και πρέπει να εφαρμόζονται και οι νόμοι. Και βεβαίως σε κάθε περίπτωση ο πελάτης έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, μπορεί να υπαγορεύει τους όρους του από αυτόν ο οποίος λαμβάνει μία σύμβαση για τον τρόπο με τον οποίο θα την εκπληρώσει αλλά και για κώδικε συμπεριφορά. Επίση μπορούν να βοηθούν οι πελάτε με το να απευθύνονται σε ηθικέ εταιρείε, ακόμα και αν αυτέ οι εταιρείε δεν κάνουν χαμηλότερη προσφορά. Επίση μπορούν οι πελάτε να τονίσουν την ε, σημασία του να ανήκει μια εταιρεία σε μια ένωση η οποία έχει κάποιε προδιαγραφέ όπω η δική μα ένωση. Θα ήθελα τώρα να σα αναφέρω κάποιε σκέψει για το πού μπορεί να πάει αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι σε μια θέση κλειδί καθώς μπορεί να τονίσει στα κράτη μέλη τη σημασία της σωστής ρύθμισης αυτού του κλάδου. Αυτή τη στιγμή ο κοινό μας εχθρός είναι η αδράνεια. Οι κανόνες και οι νόμοι που υπάρχουν στα χαρτιά πρέπει να ξεκαθαρίσουν εκεί όπου δεν είναι σαφείς και να εφαρμόζονται εκεί που δεν εφαρμόζονται. Επίσης ο κλάδος Βεβαίω θέλει να λάβει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Θέλει ο ιδιωτικό τομέα ξεκάθαρου κανόνε. συγκρίζει ζώνες απλά περιπλέκουν την σωστή παροχή υπηρεσιών σε αυτούς που τις χρειάζονται. Στο άλλο άκρο του φάσματος επίσης είναι εξίσου σημαντικό ο κλάδος να μην ρυθμιστεί τόσο ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει ή να τις βάλουμε αν θέλετε έναν ζουρλομανδία έτσι ώστε να μην μπορεί να συνεχίσει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ειρήνης και σταθερότητας. Μπορεί βεβαίω αυτά κάποιου να τους χαροποιούν, στην πραγματικότητα θα αποτελέσουν πύριο νίκη και αυτοί οι οποίοι θα χάσουν τελικά θα είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στι ε, συγκρούσει και βασίζονται στον ιδιωτικό τομέα για τι επιχειρήσει ειρήνη και σταθερότητα για να ξαναχτιστούν αυτές οι καταστραμμένες κοινωνίες. Ο ιδιωτικός τομέας ε, έχει υποστεί την κριτική βεβαίως στο παρελθόν, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα και επαγγελματισμό που φέρνει σε αυτέ τι επιχειρήσει και οτιδήποτε καθιστά τι ειρηνευτικές επιχειρήσει καλύτερε και πιο αποτελεσματικέ οπωσδήποτε είναι θετικό. Όπω είπα στην αρχή όλοι οι ανθρωπιστέ είμαστε και έχουμε έναν κοινό στόχο. Επιτυχεί ειρηνευτικέ επιχειρήσει που θα φέρουν σταθερή ειρήνη και ασφάλεια στις κοινωνίες τις ρημαγμένες από τον πόλεμο. Και εμείς αποτελούμε έναν ηθικό εταίρο σε αυτό το στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μεσνέρ. Ωραία, καταλάβαμε πολύ καλά ότι οι υπηρεσίε ασφαλεία, οι ιδιωτικέ υπηρεσίε ασφαλεία, οι ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία και ιδιωτικέ στρατιωτικέ εταιρείε αποτελούν ένα ευημερούντα τομέα, ένα τομέα που ανθεί. Ε, και υφίσταται ήδη μια ρύθμιση, αν καταλάβαμε καλά ε, δεν ξέρω, αλλά κάπως ε, μου προκάλεσαν κάποια σύγχυση παρουσιάσεις και δεν, μας, ε, και δεν με έπεισαν πλήρως. Κύριε Κολανόφσκι, εργάζεστε για τον Ερθρό Σταυρό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ που καλέσατε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερθρού Σταυρού για να λάβει μέρος σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εγώ θα σεβαστώ τα 10 λεπτά του χρόνου ομιλία, αλλά θα ήθελα προηγουμένω να σχολιάσω τα όσα είπε ο κ. Μέσνερ. Όταν λέτε ότι είμαστε όλοι ανθρωπιστές, ε, θα πρέπει να πω ότι διαφωνώ μαζί σα Ή τουλάχιστον ο δικός μας ορισμός ε, είναι διαφορετικό από το δικό σα. Τώρα θα επανέλθω στην παρουσίασή μου για το Διεθνές ε, Ανθρωπιστικό Δίκαιο και για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκ μέρου των ιδιωτικών εταιρείων ασφαλεία και ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών η παρουσία αυτών των εταιριών σε δάφιο που υπάρχουν ένοπλε σειράξει ή άλλα φαινόμενα εσωτερική βία, δεν συνιστούν ε, καινοφανέ φαινόμενο. Αλλά θεωρώ ότι ο αριθμό του, τουλάχιστον όσον αφορά το προσωπικό τους και τις των δραστηριοτήτων του, εξελίχθηκαν πάρα πολύ τα τελευταία αυτά χρόνια. Οι ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία και ιδιωτικέ στρατιωτικέ εταιρείε δεν μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω η ονομασία που του δίνουμε. Αν δούμε το διεθνέ ε, δίκαιο, ε, επικεντρώνεται στις βασικές τους δραστηριότητες, δηλαδή εμπλέκονται σε δραστηριότητες που προσεγγίζουν την καρδιά, θα λέγαμε, των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Ακούσαμε κατά επανάληψη και το ακούσαμε και εδώ προηγουμένω ότι οι εταιρίες εταιρείες ασφαλείας και οι δυτικές στρατιωτικές λειτουργούν σε ένα είδος νομικού φλού, νομικής ασάφειας. Ε, αυτό είναι εν μέρη αληθές και δεν διευκρινίζει το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας. Υπάρχει το θέμα της ατιμορρησίας ε, και πολλά τέτοια παραδείγματα αναφέρονται και στον τύπο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα διτό πρόβλημα. Η δικαιοδοτική αρμοδιότητα των χωρών, όχι, όλων, όχι όλων, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν δικαιοδοτική αρμοδιότητα και η δυσκολία από την άλλη να διεξαχθεί μια έρευνα στο πλαίσιο, για παράδειγμα, μια ένοπλη σύραξη. Πόσο μάλλον ε, ε, σε σχέση με κάποιους νομικούς κανόνες που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Είναι Προφανές ότι, για παράδειγμα, στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι δυνατόν βάσει αυτού του δικαίου να κρίνει κανείς ε, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ακόμα και σε χώρες όπως η Γαλλία ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια όσον αφορά τη διενέργεια μιας έρευνας σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ένοπλες ε, σειράξει. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι οι ίδιες ε, οι χώρες ε, να αποφανθούν για αυτές τις ε, πράξεις δεν είναι οι χώρες από τις οποίες προέρχονται τα μέλη αυτών των ιδιωτικών εταιριών αλλά οι χώρες όπου δρούν αυτές οι εταιρείες. Αλλά όπως σας είπα στις χώρες αυτές υπάρχουν ένοπλες σειράξεις και όπου τα δικαιοδοτικά όργανα έχουν αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και υπάρχουν τεράστια προβλήματα πρακτικής φύσεως σε σχέση με αυτή την αναστάτωση σε αυτές τις περιοχές. Παρατηρούμε επίσης, και αυτό είναι ιδιαίτερος λυπηρό, ότι ορισμένες εταιρείε ε, ε, χαίρουν ατιμορρησίες βάσει μιας διμερούς συμφωνίας. Για παράδειγμα, ε, μια State Force Agreement, μια συμφωνία ή στο πλαίσιο ε, πολυεθνικών επιχειρήσεων που επεκτείνονται επίσης και στους πολίτες που συνοδεύουν αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Τώρα, ας έρθουμε σε κάποια νομικά ζητήματα εις βάθος νομικά ζητήματα. Η Ελβετία μαζί με τον Ερθρό Σταυρό ε, ανέλαβε μια πρωτοβουλία σε σχέση με το ζήτημα των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας. Έχουμε εδώ το σχετικό έγγραφο. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας δεν είναι βεβαίως να νομοποιηθούν ή να ποινικοποιηθούν οι εταιρείε αυτές, αλλά να εξετάσουμε εις βάθος αυτή την προβληματική. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να συζητήσουμε για τις υποχρεώσεις που προέρχονται από το διεθνές δίκαιο και θα πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητε αυτών των εταιριών και που ορίζουν τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι διάφορες χώρες για να προωθήσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, έξι χώρες μέλη συμμετείχαν στην ε, πρωτοβουλία αυτή, 17 χώρες συνολικά. Και επίσης ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας βεβαίως και ιδιωτικές αρνητικές εταιρείες συμμετείχαν καθώς και πρόσωποι του, Think Tank, ε, διάφορες ακαδημίες κλπ. Η πρωτοβουλία κατέληξε αυτή σε αυτό το έγγραφο του Μοντρέ που επισημαίνει τις διάφορες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο αυτό και που παρέχει έναν κατάλογο των σωστών ε, πρακτικών, κάτι το οποίο ανέφερε ο κ. Κίνησε και ο κ. Μέσνε και που θα πρέπει, ε, μπορούν ε, και στο έγγραφο αυτό, μπορούν στο κείμενο αυτό του Μοντρέ, μπορούν να προσφύγουν οι χώρες μέλη. Δεν, είναι, δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο αυτό υπενθυμίζει ότι οι χώρες δεν μπορούν να απαλλαγούν από τις δικές τους υποχρεώσεις προσλαμβάνοντας μια ιδιωτική εταιρεία ή κάνοντας ένα συμβόλαιο μια ιδιωτική εταιρεία έχουν κάποιες υποχρεώσεις των οποίων η εμβέλεια ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις. Επίσης, το έγγραφο λέει ότι υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες που οι χώρες μέλη δεν είναι δυνατόν να θέσουν σε τέτοιε εταιρείε. Για παράδειγμα, την ε, άσκηση ε, ε, τα καθήκοντα ενός αξιωματικού για παράδειγμα. Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι η χώρα θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και βλέπουμε ότι όλες οι χώρες μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης που αφορά ακριβώς το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υιοθετώντα κάποια μέτρα που έχουν στόχο την ε, καλύτερη παρακολούθηση των παραβιάσεων και το ίδιο ισχύει και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μέρη να αναρθούν αποζημιώσει στα θύματα. Επίση, υπενθυμίζει ότι οι χώρε είναι άμεσα υπεύθυνε για τη συμπεριφορά των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας, ιδιωτικών στρατικών εταιρείες, ε, ε, εταιριών συγγνώμη, που λογοδοτούν στις χώρες μέλη, αυτή τη στιγμή ε, συμμετέχουν στα κανονικά στατεύματα αυτής της χώρας ή που εξοδοτούνται από τις χώρες μέλη να εκπληρώσουν ορισμένα καθήκοντα. Τώρα όσον αφορά το στάτους αυτών των ιδιωτικών εταιριών και το στάτους, το καθεστώς του προσωπικού τους, διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να θεωρηθούν πολίτες σε σχέση με το διεθνές ανθρωπαστικό δικαίο, αλλά χάνουν την προστασία αυτή που χορηγείται στους πολίτες εφόσον λάβουν μέρος σε εχθροπρεξίες. Και το ίδιο οι υπάλληλοι αυτών των εταιριών θα πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και είναι ποινικά υπόλογοι για τυχόν παραβιάσεις. Πέρα από αυτές τις νομικές σκέψεις, το κείμενο του Μαντρέ προτείνει ένα κατάλογο 70 ορθών πρακτικών για να καθοδηγεί τις χώρες που θέλουν να εκπληρώσουν σωστά τις δικές τους υποχρώσεις. Μεταξύ αυτών των πρακτικών έχουμε την, ε, ένα σύστημα χορήγησης αδειών Επίσης μια σωστή ρύθμιση για αυτές τις ιδιωτικές εταιρείε ασφαλείας, το οποίο ε, σημαίνει ότι κάθε χώρας μέλη θα πρέπει να εξετάζει το παρελθόν αυτών των εταιριών ασφαλείας. Επίσης θέματα ε, δικαιοδοτικής ε, αρμοδιότητας κλπ. Θα πρέπει επίσης να πετούνται από αυτές τις εταιρείες σωστές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού σωστή κατάρτιση του προσωπικού σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Επίσης, ε, σωστές ε, διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή ε, μιλάμε για τη χρήση βίας. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια εσωτερική πειθαρχία στις εταιρείε αυτές. και επίσης εδώ στο έγγραφο έχουμε συνημένο ένα έγγραφο του κυρίου Μέστρο που αναφέρει ακριβώς αυτές, αυτό τον κατάλογο των σωστών πρακτικών. Ε, το Συμβούλιο των Εθνών διαφέρθηκε για αυτή την πρωτοβουλία του Ερυθρού Σταυρού και έγινε μια ακρόαση με το ελβετικό τμήμα ε, σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή. Ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε μέλη μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να καταπολεμήσουν αυτό το αδικαιολόγητο αίσθημα ατιμορρησία εκ μέρου των ιδιωτικών εταιριών. Αναγνωρίζοντα τη χρησιμότητα του εγγράφου του Μαντρέ και αναφέροντα το έγγραφο αυτό στι συζητήσει του με τρίτε χώρε, καθώ και με τι ιδιωτικέ εταιρείε, με τι ίδιε ιδιωτικέ εταιρείε, κάτι το οποίο θα ήταν ένα καλό παράδειγμα εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πρόθεση του σεβασμού του ανθρωπιστικού δικαίου θα ήθελα ο κατάλογο των καλών πρακτικών πραγματικά να εμπνεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε μέλη στι προσπάθειέ του να προλάβουν τι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτω ώστε να καταπολεμήσουν καλύτερα αυτά τα φαινόμενα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Παίζω λίγο με τα μικρόφωνα το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα μπορούσαν να πάρουν το λόγο. Υπάρχει κάποιο από το Συμβούλιο που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι. Κύριο Κύριος Κίνγκ. Ευχαριστώ και πολύ σύντομα. Το θέμα της ρύθμιση αυτών των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως η Κομισιόν γνωρίζει τη σημασία αυτού του θέματο. Εμείς ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέτουμε τέτοια θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, απέναντι στις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα του Ιράκ και του Αφγανιστάν δημιουργούν, θέτουν δύσκολα ερωτήματα το πώς θα διώξουμε αυτές τις εταιρείες για να μην υπάρξει ατιμορρησία. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που λένε ότι οι κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου ισχύουν και για τα κράτη και για τους υπόλοιπους φορείς και υπάρχει και ατομική ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση, ε, είτε την παραβίαση την έχει κάνει η κράτο, είτε ιδιωτικό φορέα ή οποιοδήποτε άλλο φορέα. Ε, υπάρχει αυτό το κείμενο του Μοντρέ που είναι ένα καλό βήμα προ τα εμπρό. Ε, προωθεί το ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνέ δίκαιο, αλλά αυτό το κείμενο υιοθετήθηκε πρόσφατα και η πρόκληση τώρα είναι να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του. Η Κομισιόν θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, η Κομισιόν σημειώνει τη σημασία της ε, επίβλεψης των ιδιωτικών εταιριών ε, και αυτό το αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας του 2006. Σας ευχαριστώ την προσοχή σε ένα πρόγραμμα που υποστήριξε η Κομισιόν για αυτό το θέμα, που είναι ένα πρόγραμμα ε, για την Νότια Ευρώπη, που οδήγησε στο κώδικα διοντολογίας του Σαράγεβο για τον έλεγχο των μικρών όπλων. Εκεί έχουμε βασικά πρότυπα για τον επαγγελματισμό και την παροχή υπηρεσιών από όλο το προσωπικό και τις εταιρείε αυτές, τις ιδιωτικές. Ο κώδικας διοντολογίας καλύπτει διάφορες, διάφορες τομείς, την επιλογή του προσωπικού, την κατάρτισή του, ε, μη διάκριση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τους με τους πελάτες, ε, την αστυνομία και τις υπόλοιπε εταιρείε. Ε, Επίσης, ε, για τις ε, Υπάρχουν τέτοιοι κανόνες για τις προμήθειες, για την ποιότητα των υπηρεσιών, το επίπεδο κατάρτισης και το σεβασμό της εθνικής νομοθεσίας. Ε, αυτός είναι θελοντικός κώδικας διοντολογία. Η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό και τον τρόπο εφαρμογή του. Ευχαριστώ κύριο Γκαλέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο άκουσα όσο το άκουσα ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Το έγγραφο του Μοντρέ δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά από αυτά τα οποία ακούγονται νομίζω ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε ανεπιφύλακτα. Για το θέμα αυτό, για τις ιδιωτικές εταιρείε ασφαλείας και στρατιωτικές εταιρείε δεν πρέπει να υπάρχουν χώροι χωρίς δίκαιο στις χώρες δηλαδή όπου επεμβαίνουν αυτές οι εταιρείες μέσω της επέμβασής τους να μην δημιουργείται μια σφαίρα η οποία είναι εις βάρος των ανθρώπων εκεί πέρα. Αν δούμε τις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας υπό κανονικές συνθήκες προστατεύουν είτε αντικείμενα είτε πρόσωπα. Ένα αντικείμενο Εντάξει, προφανώς είναι περιφραγμένο και έχει κάποιες διαστάσεις όσον αφορά δε τα πρόσωπα κινούνται μαζί με το πρόσωπο και μαζί κινείται και ο τομέας αρμοδιότητάς τους. Για μένα λοιπόν είναι ζήτημα φυσιολογικής ε, της απλής νομοθεσίας της εκάστοτε χώρας το ποιες αρμοδιότητες έχουν αυτές οι εταιρείε εάν ε, οπλοφορούν ή όχι κατά κανόνα μπορεί αυτό να συμβαίνει, αλλά δεν είναι κάποιος χώρος χωρίς ε, δίκαιο που δημιουργείται από την επέμβαση αυτών των εταιριών. Γι' αυτό πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιώ επικούς της ίδιας χώρας ή αλλοδαπούς σε αυτό τον τομέα. Και για τους δύο πρέπει να ισχύει το ίδιο δίκαιο. Καμία κυβέρνηση δεν θα διευκολύνει νομίζω το έργο τους με το να προσλαμβάνει ανθρώπους ε, για κάποιες αποστολές τις οποίες τελικά πρέπει να τις κάνει ίδια. Για τον τομέα των ιδιωτικών εταιριών ασφαλείας ε, δεν είναι νομίζω ναι, είναι ζήτημα κάποιες κυβέρνησης, ε, είναι μάλλον κάποια εταιρεία που προσλαμβάνει αυτές τις εταιρείες. Όσον αφορά τις ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες, οι άνθρωποι αυτοί είναι μισθοφόροι χρήματα παίρνουν γι' αυτό και εκεί όταν τους προσλαμβάνει μια κυβέρνηση που έχει το δικαίωμα όταν δεν είναι σε θέση μόνη της με το δικό της στρατό να διασφαλίσει την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της χώρας αλλά και εκεί πέρα δεν θα επιτρέπεται αυτό να είναι πρόσχημα για ένα κράτος ή μια κυβέρνηση να, επιτρέψει, να επιτρέπει να ισχύει διαφορετικό δίκαιο από ό,τι για το δικό του στρατό. Και οπωσδήποτε ε, δεν μπορεί μια κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να αποφύγει τις διεθνείς υποχρεώσεις της. Αυτό πρέπει να είναι το μέτρο νομίζω. Και να το δούμε μετά συγκεκριμένα και να δούμε πού υπάρχουν αυτές οι εγγυήσεις ε, και πού όχι. Και αναλόγως να ακούω πω η Κομισιόν δεν είναι αρμόδια οπότε είναι ζήτημα των κρατών μελών κάθε κράτος μέλος μετά να φροντίσει τα σχετικά και να προσέχει το πως ε, δρά. Επίσης όταν μιλάμε για διμερείς ε, συμφωνίες, αν γίνεται πύχη κάτι και συμφωνείτε κάτι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, έτσι ώστε στρατιώτες μας να προστατεύονται π.χ. από μια ιδιωτική εταιρεία, τότε αυτό από τη δική μας σκοπιά δεν πρέπει να σημαίνει ότι ε, συμφωνούμε σε κάτι χωρίς ε, συνέπειες, χωρίς να υπάρχουν συνέπειες, γιατί ανοίγουμε διάπλατη την πόρτα για κατάχρηση μετά και του διεθνούς ε, δικαίου μέσω της ε, τεθλασμένης ε, αυτών των ιδιωτικών στρατιωτικών εταιριών και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Γκαλέ. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο, άλλος βουλευτής. Όχι. Δεν μιλήσατε για την ομάδα εργασία του ΟΗΕ για του μισθοφόρου. Τι γνώμη έχετε για τη δουλειά που κάνει, για την έρευνα που κάνει, για τις συστάσεις που δίνει. Ποιο εμπλέκεται σε αυτές τι δραστηριότητε, Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, θέλω να πω ότι είχαμε ε, καλέσει τον πρόεδρο τη ομάδα εργασία του ΟΗΕ για του μισθοφόρου, αλλά δεν μπορούσε να έρθει δυστυχώ ε, γιατί είχε κάποιε υποχρεώσει σήμερα. Το συναντήσαμε στη Γενέβη. Και μετά από αυτή τη συνάντηση, μάλιστα με την ομάδα εργασία του ΟΗΕ, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τη σημερινή ακρόαση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είπε ο κύριο Γκαλέρ, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι στις, επιχειρη... στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις ε, σε όλες τις επιχειρήσεις που αφορούν την ε, ασφάλεια και την άμυνα, τα θέματα τα ανθρωπιστικά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θα πρέπει να υπάρχει ένας αξιωματικός συνδέσμο ίσως ε, μεταξύ της ευρωπαϊκής επιχείρησης και των εταιριών, αυτών των ιδιωτικών εταιριών που δίνουν αυτές τις υπηρεσίες βοηθώντας ίσως ε, στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Θα πρέπει να υπάρχει ένας συστηματικός σύνδεσμος, ε, ούτως ώστε να υπάρχει ε, εστίαση στο σεβάσμα των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και στο ανθρωπιστικό δίκαιο, για να μην γινόμαστε μάρτυρες σοβαρότητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι πολύ πιο πολλοί άριθμες από αυτές που είπατε κύριε Κίνση και κύριε Μέσνερ. Εσείς κύριε Κίνση αναφέρατε μέρος γνωστές περιπτώσει πιο πρόσφατες και λιγότερο πρόσφατες. Ο κίνδυνος είναι ότι στην υπεργολαβία, στην αλυσίδα υπεργολαβίες διαφόρων αποστολών ε, κατά τη διάρκεια πολέμων ή μετά τους πολέμους στα πλαίσια μια σχέσης με τους ντόπιου πληθυσμού που είναι ευπαθείς, που δυσκολεύονται εκεί θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και η υπεργολαβή ορισμένων δραστηριοτήτων, γιατί ο κ. Κολανόφσκι υπενθύμησε ότι όλε οι δραστηριότητε δεν μπορούν να δοθούν σε υπεργολάβου. Δεν θα πρέπει λοιπόν όταν, δίνουμε, όταν δίδονται κάποιε δραστηριότητε υπεργολάβου να λησμονούνται οι ευθύνε που έχει ο ανάδοχο και βέβαια θα πρέπει να λησμονά και το κράτο ε, τι ευθύνε που έχει σε αυτόν τον τομέα. Για αυτή την ομάδα του ΟΗΕ που δουλεύει για τους μισθοφόρους θα ήθελε κάποιος να πάρει τον λόγο. Να μας πει ποια είναι η εκτίμησή του για τη δουλειά που κάνει αυτή η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ. Και κύριε Κολονάφη, να μας πείτε, αν ξέρετε, τι προοπτικές υπάρχουν. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2008 έγινε μια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ με την με την ε, συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών της ε, Ελβετικής Κυβέρνησης και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Προσπάθησαν να ανταλλάξουν απόψεις για κάποια νομικά θέματα και να δώσουν ε, την άποψή τους για τεχνικά θέματα. Συνεχίζεται η δουλειά από ό,τι ξέρω και δεν νομίζω ότι απόκειται σε εμά να σχολιάσουμε σε αυτή τη φάση τη δουλειά που γίνεται ως Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού. Αλλά υπάρχει ο διάλογο. συνεχίζεται ο διάλογο. Ελπίζουμε ότι κάπου θα καταλήξει. Όπω είπε και ο κύριο Σκίνση, έχουμε αυτόν τον ορισμό του μισθοφόρου που δεν καλύπτει ικανοποιητικά τι ε, ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλείας. Ο ορισμός του μισθοφόρου στο διεθνές δίκαιο είναι τόσο περιοριστικός που ελάχιστοι καλύπτονται ε, και εντάσσονται ε, σε αυτόν τον ορισμό. Κύριε Κίνσνε, ναι, κύριε, κύριε να προσθέσετε κάτι στον, ε, στη συζήτηση. Εγώ μίλησα σε αυτή την Επιτροπή για το θέμα των μισθοφόρων και των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας. Είναι καλή δουλειά που γίνεται σε αυτήν την ομάδα εργασία. Προσπαθούν να κάνουν μια διάκριση ανάμεσα στου μισθοφόρου που είναι παράνομοι ε, σε μάχες και σε πολέμους και στις επιχειρήσεις των ιδιωτικών εταιριών ασφάλειας. Ίσως υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει μαζί με τον ΟΗΕ σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει κανονισμού. Εκεί μπορούμε να έχουμε επιτυχία. Πιο πολύ παρά στον ΟΗΕ. Αλλά και οι δύο οργανισμοί θα πρέπει να δουλέψουν ε, εκ παραλίλου. Πάντως πιστεύω ότι ο κανονισμός θα περάσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ΟΗΕ. Γιατί έχουμε αυτή τη διεθνή σύμβαση σε επίπεδο ΟΗΕ για που απαγορεύει την στρατολόγηση, χρήση και χρηματοδότηση κτλ η οποία δεν δούλεψε. Στο έγγραφό μου ε, λέω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουν και οι δύο οργανισμοί να προωθήσουν μια διεθνή σύμβαση που θα ρυθμίσει τις δραστηριότητε των ιδιωτικών εταιριών. Καταρχάς όμως πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει πολλά σε αυτό το τομέα, να ρυθμίσει τις δραστηριότητες ε, ε, των εταιριών αυτών. Επίσης, οι ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο επιτρέπει ε, στις ε, εταιρείε αυτές να κινούνται από χώρα σε χώρα. Αν μια εθνική νομοθεσία είναι πολύ περιοριστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάει σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ε, καλό θα ήταν λοιπόν να κινηθούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να εμποδίσουμε αυτέ τι εταιρείε να παρακάμπτουν την, νομοθε... την εθνική νομοθεσία μετακινούμενε σε άλλο κράτο μέλο. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να πω λίγα γρήγορα όσον αφορά την ομάδα εργασία των Ηνωμένων Εθνών. Και εγώ έχω μιλήσει εντόπιον αυτή τη ομάδα και πραγματικά κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά σε σχέση με το θέμα αυτό. Η ομάδα εργασία ξεκίνησε ω ε, ειδικό συγητή σε Ηνωμένα Έθνη για το θέμα των μισθοφόρων και στη συνέχεια εξελίσσεται στη σημερινή τη μορφή. Εάν ε, η Υποεπιτροπή ενδιαφέρεται να συνομιλήσει με την ομάδα εργασία, πραγματικά θα ήθελα να σας στήσω τον Αλεξάνδρ Ακίτον που είναι, από τη Ρωσία που είναι συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας και είναι πραγματικά εξαίρετος ε, στην ιδιότητά του αυτή. Ένα άλλο μέλος της ομάδας εργασίας είναι ένας προηγούμενος ειδικό εισηγητής, ο Dr. Σάστρη Σιμίν από το Φίτζι, ο οποίος είναι ένας, διεθνή, ένας εμπειρογνώμων για το θέμα αυτό και πραγματικά είναι σε θέση να γνωμοδοτήσει με ξέρετο τρόπο ενώπιον τη επιτροπή. Οι σχέσει μας υπήρχαν αρκετά καλές μέχρι στιγμή. Δυστυχώ, το γεγονός ότι η ομάδα εργασία επικεντρώνει την προσοχή τη στου μισθοφόρου. και όχι στην εταιρεία για την, στις εταιρείες στις οποίες αναφερόμαστε σήμερα έχει επιβραδύνει κάπως την πρόοδο των εργασιών. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον επίπεδο της ομάδας εργασίας γιατί ακριβώς περιορίζεται η δουλειά τους λόγω ακριβώς της συγκεκριμένης αποστολής τους να ασχοληθούν με το θέμα των μισθοφόρων αντί ε, και νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ανανέωση της εντολής τους από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτως ώστε να επεκταθεί. Ευχαριστούμε πολύ και εδώ θα ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση που εφόσον τα μέλη το επιθυμούν θα μπορέσουν να έρθουν ε, σε επαφή με αυτή την ομάδα εργασίας και να υπάρξει μια συνέχεια υπό τη μορφή της σύνταξη μιας έκθεσης πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να συνεχίσουμε ε, τις εργασίες μας με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 4 ε, της ημερήσιας διάταξης παρουσίας εκ μέρους του κυρίου Evans για το θέμα της ελευθερία της ε, θρησκείας ένα θέμα το οποίο έχουμε προσεγγίσει κατά επανάληψη στο επίπεδο αυτής της Επιτροπής. Είχαμε καλέσει την κυρία Ασμά Ονζή ε, στις 10 Ιουνίου και επίσης και στην ε, Γενέβη. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί κατά επανάληψη ε, με το οποίο ασχολείται και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και υπάρχει ένα σχετικής, ο σχετικός ε, είναι ένα θέμα το οποίο έχει μια πολιτική βαρύτητα και το οποίο έχει δώσει ένα τόσο πολλές συζητήσεις όσον αφορά την Ευρωμεσογειακή Ένωση ε, ήδη από την εποχή που είχαν δημοσιευθεί τα σκίτσα του Μωάμεθ. Ε, θα θυμάστε ότι από την εποχή εκείνη αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνας του κυρίου εγώ είμαι συγγήτρια για μια έκθεση με το θέμα αυτό στην... Ε, Ευρωμεσογειακή Συνέλευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την μελέτη σήμερα. Όπως θα ακούσατε, δεν χρειάζονται πολλά λόγια εκ μέρους μου για να σας πω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό. Και ε, ε, δεν θα ήθελα να το επισημάνω άλλη μια φορά. Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω ωστόσο είναι ότι αυτό το ειδικό θέμα της ε, ελευθερίας των θρησκευτικών πεπιθήσεων και της ελευθερίας της έκφρασης παρόλο που είναι πραγματικά ένα θέμα αυτό καθ' αυτό νομίζω από την άλλη θα πρέπει να προσλαμβάνεται ως τμήμα ενός ευρύτερου πλαισίου και είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε το ειδικό αυτό θέμα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Και εγώ από την πλευρά μου πιστεύω ότι αυτό το γενικότερο πλαίσιο αποτελεί τμήμα μιας ακόμα πιο πλατιάς συζήτησης ε, που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή και αφορά την σωστή θέση και τον ρόλο των συστημάτων θρησκευτικών πεπιθήσεων στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες εν γέννη και στην, ε, στο χώρο της κοινή γνώμης ιδιαίτερα. Και βεβαίω ε, υπήρξαν διάφορες εκδηλώσεις αυτής της πλατιάς συζήτησης και νομίζω ότι εδώ ασχολούμεθα με μια διάσταση αυτού του θέματος σε σχέση με το ζήτημα της ελευθερίας θρησκευτική ε, έκφρασης. Αλλά υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που αφορούν για παράδειγμα τα θρησκευτικά σύμβολα, ε, την ε, δυνατότητα ρύθμισης όσον αφορά διαδικασίε πρόσληψη βάσει θρησκευτικών πεπιθήσεων κλπ. Είναι θέματα τα οποία συναρτώνται στενά μεταξύ τους. Και Μία από τι προσεγγίσει αυτή τη έκθεση αφορά την ειδική σχέση αλληλεπίδραση μεταξύ θρησκευτική ε, πεποίθηση και ελεύθερη έκφραση, ε, Δύο πλατύτερα θέματα, τα οποία θα πρέπει να λησμονούμε. Το δεύτερο γενικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να αναφέρω σε σχέση με αυτή την έκθεση, είναι το εξή. Αναπόφευκτα η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στη μία προσέγγιση του θέματος από την προοπτική του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και ε, Βεβαίω αυτό θα ανέμενε κανεί από μια έκθεση αυτή τη Επιτροπή. Ε, Επίση είναι σημαντικό να γνωρίσουμε άλλη μια φορά ότι υπάρχουν και άλλες προπτικέ που αφορούν την, το θέμα αυτό από μια πλατύτερη κοινωνιολογική άποψη. Εγώ θα επισέλθω σε αυτό το θέμα, αλλά βεβαίως θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι υπάρχουν κοινωνιολογικές, θεολογικές κλπ. διαστάσεις όταν ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά και που δεν θα πρέπει να τις βάζουμε στην άκρη. Τώρα, αν γυρίσουμε σε την έκθεση, θα ήθελα να πω ότι η έκθεση αυτή είναι σχετικά βραχία σε σχέση με κάποια θέματα που ορισμένοι θα ήθελαν ίσως να δουν να αναφέρονται διαμακρών. Για παράδειγμα, όσον αφορά μια αριστική απάντηση στο θέμα που θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς μια ισορροπία μεταξύ των ε, φόβων αυτών. Η απάντηση που προσπαθούμε να προωθήσουμε είναι ότι αυτός είναι ένας εσφαλμένος τρόπος προσέγγισης αυτού του θέματος αυτό το οποίο κάνει η έρευνα, η μελέτη, προσπαθεί να σκεγγραφίσει αυτό που πιστεύω ότι είναι ένας πιο νέος τρόπος προσέγγισης αυτού του θέματος με όρους που προσπαθεί να θέσει μια πρόκληση στους ε, παλιότερους όρους με τους οποίους συνήθως πραγματεύονται το θέμα αυτό, αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Και ε, προσπαθεί από την άλλη να δώσει ε, κάποιες ε, προσεγγίσεις σε σχέση με συγκεκριμένα θέματα που ανακύπτουν. Γιατί βεβαίως δεν είναι δυνατόν να απαντήσουμε αφηρημένα τα θέματα αυτά, αλλά πάντα θα πρέπει να ασχολούμεθα με τις συγκεκριμένες ε, περιστάσεις, τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά βεβαίως είναι ουσιώδης ο τρόπος προσέγγισης αυτών των θεμάτων. Το πρώτο ουσιαστικό θέμα το οποίο θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω έχει ως εξής. Ε, κατά κάποιο τρόπο βεβαίως ε, στηρίζει όλη την έκθεση. Παρόλο που συχνά το θέμα της εξορρόπησης ε, δύο αντικρώμενων συμφερόντων, η δική μου ελευθερία θρησκευτική πεποίθησης από τη μία και η ελευθερία έκφρασης από την άλλη εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε σαν δύο αντίθετους όρους, αλλά σαν δύο συμπληρωματικές ε, πλευρές. Και κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας τα νομικά έγγραφα, δηλαδή τις αποφάσεις των δικαστηρίων, το ίδιο το κείμενο της ε, Σέμβασης και άλλων διεθνών εργαλείων. Και αυτό που στην πράξη λένε τα δικαιοδοτικά όργανα σε σχέση με αυτές τις ε, ισορροπίες. Και για να σας δώσω μια γεύση θα ήθελα να πω ότι το πρώτο σημείο κίνησης αφορά ε, ένα μια πολύ σημαντική υπόθεση όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή θρησκευτική πεποίθηση όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάθηκε ότι ο πλουραλισμός είναι αλληλένδετος με τις επιταγές μιας, δημοκρατικής, μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Αντίστοιχε διατυπώσει αναφέρονται όσον αφορά την ελευθερία τη έκφραση, όταν ο δικαστήριο λέει ότι είναι μία από τι θεμελιώδει συνιστώσει τη δημοκρατική κοινωνία και αφορά την ίδια την αυτοεκπλήρωση του ατόμου. Δηλαδή, από την άποψη της νομολογίας, η ελευθερία της ειδικής πεποίθησης, αλλά και η ελευθερία της έκφρασης θεωρούνται ίσες αξίες. Αλλά εάν επανέλθουμε στα κείμενα ε, της ίδιας της σύμβασης και των νομικών οργάνων, ε, μπορούμε να δούμε το πώς ακριβώς ε, γίνεται και θα αναφερθώ σε τρεις τρόπους, τρία παραδείγματα που αυτό γίνεται προφανές. Πρώτον, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ μορφών ε, σκέψης, ε, συνείδησης και θρησκείας και της ιδέας ότι γνώμες και ιδέες θα πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα και προστατεύονται από το άρθρο 10. Και πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε κατά πόσο κάτι αφορά, εμπίπτει στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 10. Και αυτό το οποίο συχνά λησμονούμε είναι ότι κάθε μορφή θρησκευτικής πεποίθησης που εμπίπτει στο άρθρο 9 και αλλά αυτόματα εμπίπτει, υπάγεται και στο άρθρο 10 που αφορά την ελευθερία της έκφρασης. Υπό την έννοια αυτή πρόκειται για μια πολύ στενή δομική σχέση μεταξύ των δύο. Και πάλι υπάρχει μια στενή δομική σχέση μεταξύ των δύο που επισημαίνεται όταν δούμε τι γίνεται στην πράξη. Η ιδέα ότι η έκφραση των θρησκευτικών πεπιθήσεων όπως διατυπώνεται στο άρθρο 9 ε, στην πράξη αφορά την ελευθερία της έκφρασης και το ε, δικαστήριο ξέρει ότι πράξεις που αφορούν την ελευθερία της ευθυντικής πεποίθησης τελικά εκφράζονται ελεύθερα. Η έκφραση απόψεων που δεν εκδηλώνονται από ένα που δεν είναι στο πλαίσιο ενός θρησκευτικού συστήματος, υπάρχονται ωστόσο στην προστασία του άρθρου, η συμβέλεια του άρθρου 10. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ στενή σχέση μεταξύ των δύο και είναι ξεκάθαρο όταν δούμε λεπτομερία ορισμένες από τις νομολογίες σε σχέση με τα άρθρα αυτά όταν πραγματικά βλέπουμε ότι είναι θέμα συγκυρίας ή θέμα επιλογής όταν το νομοθέτης να εστιάσει στο ένα άρθρο ή στο άλλο που η δηλαδή, την ελευθερία της κρατικής πεποίθησης την ελευθερία έκφρασης και πράγματι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη γραμμική σχέση μεταξύ της ε, ελευθερίας των σκεπτικών πεπιθύμησεων και της ελευθερίας της έκφρασης και όχι μια σχέση αντιθετική. Τώρα, όλα βέβαια αυτό το θέμα της στενής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο και τα δύο στηρίζονται, υποβαστάζονται από ένα κοινό σύστημα αξιών. Ωστόσο, από την άποψη της νομολογίας ε, υπάρχει ένα ε, περιθώριο διακριτικής ε, ευχέρειας όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τόσο το άρθρο 9 όσο και το άρθρο 10 περιγράφουν και εδώ με τον ίδιο τρόπο τους περιορισμούς θα λέγαμε όσον αφορά τα συστήματα αξιών που προσήκουν ε, στη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε σχέση με την μελλοντική τους ε, εφαρμογή. Και εδώ αναφέρομαι ε, στην εξαίρεση του άρθρου 17, το οποίο είναι ιδιαίτερως περιοριστικό και το οποίο δεν ε, ταιριάζει σε μια τέτοια σύμβαση. Εάν ε, προχωρήσουμε πέρα από αυτά τα όρια σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε σαν πιο οικείο έδαφος όσον αφορά αυτό το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση μεταξύ του τρόπου που αυτά εφαρμόζονται στην πράξη, τουλάχιστον από θεωρητική άποψη. Και το άρθρο 10 που αφορά την ελευθερία έκφρασης, εδώ διαποστώνουμε ένα αρκετά στενό περιθώριο διακριτική ευχέρεια, ενώ ε, όσον αφορά, ε, όσον αφορά τα περιθώρια εκ μέρους των ε, χωρών. Ενώ δεν ισχύει το ίδιο για, το, για την ελευθερία θρησκευτικών πεπιθήσεων, όπου το περιθώριο αυτό είναι κάπως ευρύτερο. Και βεβαίω είναι δυνατόν να υπάρχουν διαφορετικά αποτελέσματα κάτω από διαφορετικές ε, περιστάσεις. Σε διάφορες χώρες, για παράδειγμα, Παρ' όλα αυτά υπάρχει στην πράξη μία μεγαλύτερη πιθανότητα ε, σύνθεσης ε, του αποτελέσματος σε σχέση σε συνάρτηση και με τα δύο αυτά άρθρα. Και στα λίγα λεπτά που μου απομένουν θα ήθελα να σας πω το εξής. Ε, το δικαστήριο ε, καλεί τα δικαστήρια να αποφανθούν με έναν ουδέτερο τρόπο όσον αφορά θρησκευτικές και μη θρησκευτικές πεπιθήσεις. Δηλαδή οι χώρες δεν δίνουν μια προτεραιότητα στην ελευθερία της πεποίθησης έναντι, δεν δίνουν μια προτεραιότητα έναντι άλλων μορφών πεποίθησης, αλλά καλούνται να είναι αμερόληπτοι στον τρόπο που προσεγγίζουν αυτά τα θέματα. Και είναι σημαντικό όμως να θέσουμε αυτά, αυτές τις αξίες παράλληλα με κάποιες άλλες αξίες. Για παράδειγμα την ενίσχυση της ανεξιθρησκείας και του πλουραλισμού. Αυτό δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα της προστασίας αυτών των αξιών, αλλά συνιστά ένα θετικό στόχο ο οποίος πρέπει να εκπληρώνεται. Δηλαδή, οι πιστοί και μη πιστοί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ένα υψηλό επίπεδο προκλήσεων σε σχέση με τις θρησκευτικέ αξίες από τη μία και την ανεξιθρησκεία από την άλλη. Και καθήκον των χωρών είναι να απολαμβάνουν, τόσο οι πιστοί όσο και οι μη πιστοί, ε, απολαμβάνουν των ίδιων ε, δικαιωμάτων. Και μόνον εφόσον ο τρόπος με τον οποίο εκφράζονται κάποιες αξίες ε, παραβιάζει το πνεύμα ανεξιθρησκείας με έναν κακόβουλο τρόπο θα πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος από την προοπτική της ανεξιθρησκείας. Τέλος, υπάρχει η ανάγκη προστασίας των ελευθεριών των άλλων. Και εδώ η έννοια κλειδί είναι η αρχή του σεβασμού. Η έννοια του σεβασμού είναι μία από τις αρχές, από τις αξίες ε, κλειδιά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 Πρέπει να σεβόμαστε βεβαίω και τα μικρόφωνα, εκτό των άλλων. Φαίνεται πως έχω κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα με την αρχή του, του σεβασμού. Το τρίτο λοιπόν από αυτά τα βασικά ζητήματα είναι η αρχή του σεβασμού των διαφόρων απόψεων. Και πάλι το δικαστήριο στην ομολογία του πολλές φορές έχει τονίσει πως ίσως χρειάζονται περιορισμοί και στις δύο ελευθερίες για να συμβιβαστούν τα συμφέροντα διαφόρων ομάδων και να γίνονται σεβαστές οι, τα πιστεύω όλων. Αυτό το οποίο λοιπόν μπορούμε να πούμε συμπερασματικά είναι πως αυτό το οποίο έχουμε και αναφέρει σε πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια η έκθεση είναι πως μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τη σχέση ανάμεσα στην ε, θρησκευτική ελευθερία και την ε, ελευθερία έκφρασης με κάπως διαφορετικό τρόπο, με μια σύνθεση ανάμεσα στα δύο, με το σεβασμό των ιδεών και των απόψεων σε ένα κοινό φάσμα που βεβαίως ε, όλες υποστηρίζονται από κοινέ αρχές και από την κοινή προσέγγιση της ουδετερότητας, της αμεροληψίας, του πλουραλισμού, της ανεκτικότητας και του σεβασμού στο πώς ε, εκδιπλώνονται σε συγκεκριμένες ε, περιστάσεις. Μπορεί βεβαίως κάποιος να πει πως ωραία είναι όλα αυτά, αλλά πολύ ομιχλώδη. Τι γίνεται στην πράξη. Κοιτάξτε, αν, είναι, αν παίρναμε συγκεκριμένες μεμονωμένες ε, περιπτώσεις, μπορούμε να δούμε πως η εφαρμογή κάθε μίας από αυτές τις αρχές μας καθοδηγεί στο να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα από το τι θα γινόταν ε, εάν απλώς κάναμε μία συζήτηση για το ποιες είναι οι πιο σημαντικές αξίες συζήτηση η οποία δυστυχώς κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται συχνότερα. Εν πάση περιπτώσει θα μείνω σε αυτά κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Εύανς. Πολύ ελκυστική είναι η παρουσίασή σας. Έχουμε την ελευθερία έκφρασης και την θρησκευτική ελευθερία. Ένας κύκλος που η μία ελευθερία εξαρτάται από την υλοποίηση της άλλης, από την ύπαρξη, την υλοποίηση της άλλης. Ε, πολύ ελκυστικό αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η ανεξιθρησκεία, ο πλουραλισμός, η ευημερία έτσι, στις κοινωνίες μας σε σχέση με τις απόψεις και τις ιδέες. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει οπισθοχώρηση και των δύο δικαιωμάτων. Δηλαδή, η θρησκευτική ελευθερία στο δημόσιο επίπεδο που αφεαυτής δεν είναι καθόλου καταδικαστέα, αλλά που θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιες εκδηλώσεις, μίσους, κάποιες ριζοσπαστικές ε, εκδηλώσεις που οδηγούν σε περιορισμού στην έκφραση, σε μείωση της ανεξιθρησκείας κτλ. Υπάρχει και περίπτωση. Λέτε ότι οι περιορισμοί που θα μπορούσαν να συμβούν για αυτές τις ελευθερίες είναι περίπου ίδιας φύσης και εξαρτώνται από την ίδια την κοινωνία και το ίδιο το κράτος. Γιατί το ίδιο το κράτος θα πρέπει να εκτιμήσει αν η άσκηση της τάδε ή της δίνα ελευθερίας, έκφρασης ή θρησκευτική ελευθερίας γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο πλουραλισμού και σεβασμού του άλλου. Αλλά μπορούμε να γίνουμε μάρτυρες ε, τεταμένων καταστάσεων, όπου μία ουδέτερη έκφραση μπορεί να προκαλέσει κάτι τρομακτικά βίαιο, όχι σε φυσικό επίπεδο κατά ανάγκη, αλλά μπορεί να προκαλέσει απίστευτες αντιδράσεις. Δηλαδή αυτός ο, ο ωραίος σας κύκλος μπορεί να αντιστραφεί. Μπορεί δηλαδή οι δύο αυτές ελευθερίες ταυτόχρονα να μειώνονται να υποσκάπτει μία την άλλη. Γίνεται αυτό. Yes, that is certainly a possibility. Ναι, είναι πράγματι μία πιθανότητα και αυτή, αλλά βεβαίω ε, όπως για όλους τους περιορισμούς μας έχει το πλαίσιο στο οποίο μιλάμε και είναι αναπόφευκτο διαφορετικές κοινωνίες ε, σε διαφορετικές στιγμές δεδομένου ε, της νομικής ε, παράδοσης τους, ε, συνταγματικής παράδοσης, των, της κατάστασης της σκεφτικής κτλ. Μπορεί να επιτύχουν αυτή την ισορροπία με διαφορετικό τρόπο υπό διαφορετικές συνθήκες. Αυτό το οποίο νομίζω είναι εξίσου σημαντικό είναι πως εάν μία λύση σε αυτές τις δυσκολίες είναι συνεχώς ένας αγώνας προς τα κάτω. Δηλαδή να πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχει ανεκτικότητα και πλουραλισμός είναι να αποκλείουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την θρησκευτική ομιλία από την δημόσια συζήτηση. Ε, το αποτέλεσμα μάλλον θα είναι το ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο την προώθηση δηλαδή της ε, συμπερίληψης των ανθρώπων και της αυτοπεποίθησής τους να εκφραστούν γενικότερα. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι οπωσδήποτε τις διάφορες εκφράσεις ε, θρησκευτικέ και μη και το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο για να διασπείρουν θρησκευτικό και εθνοτικό μίσος. Γι' αυτό δικαίως υπάρχει περιορισμός π.χ. μέσω της νομοθεσίας ε, περί ρατσιστικής ε, προπαγάνδας κτλ. Οπότε έχουμε ένα χρησιμότερο τρόπο για να περιορίσουμε τα απότατα όρια, αν θέλετε, του αποδεκτού. Εγώ αναφέρομαι στους γενικούς, αν θέλετε, περιορισμούς του πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα αντί για να δούμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα για καταστάσεις επίμαχες για το άτομο, αλλά όχι οπωσδήποτε για την ευρύτερη κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι θίξατε έναν πολύ υπαρκτό κίνδυνο, αλλά αυτό αντιμετωπίζεται με άλλο τρόπο, όπως π.χ. με την ομοθεσία, όπως σας είπα, περί ρατσιστικών δηλώσεων κτλ. Μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Αλλά και αν οποιοδήποτε άλλο θέλει να θέσει ερωτήσεις, παρακαλώ, ε, ελεύθερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι Τούρκος και θέτω και εγώ αυτό το ερώτημα που θέσατε και εσείς. Μήπως αντιστραφεί αυτός ο αγνός κύκλος και η αύξηση της θρησκευτικότητα σε μια κοινωνία να οδηγήσει σε κοινωνικές πιέσεις εκτεταμένες απέναντι σε άλλες κοινότητες ή ε, πληθυσμούς που δεν ανήκουν σε αυτή τη θρησκεία. Το θέμα είναι αν έχουμε κάποια γενή εγγύηση μέσα σε αυτό, το, αυτό το θρησκευτικό λόγο, τόσο ώστε αυτός να αναγνωρίζει την διαφορετικότητα. Είμαστε συνέχεια υποχρεωμένοι να περνάμε μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις ή η ίδια η θρησκευτικότητα μπορεί να αυτορυθμίζεται. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θέτω. Είναι δηλαδή η ικανότητα αυτορύθμισης και αυτοπεριορισμού της θρησκείας και του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ύπαρξης των άλλων ε, και ακόμα και των αντιθρησκευτικών εκδηλώσεων. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πού θα σας απαντήσει βέβαια σε αυτό ο κύριος Σέβανς. Ευχαριστώ. Το ότι μπορεί να υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου οι απόψεις που εκφράζονται δημόσια μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες σε άτομα που ανήκουν σε άλλα θρησκεύματα ή που είναι άθε να συνεχίσουν τις πρακτικές τους. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα και νομίζω ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, θα πρέπει να αποφύγουμε την εξής κατάσταση. Το να αισθανόμαστε ότι πιεζόμαστε ε, και ότι πρέπει να συμμορφωθούμε σε κάποιες σκεφτικέ πρακτικές, τις οποίες εμείς δεν πιστεύουμε. Από την άλλη δεν μπορεί να υπάρχει πραγματικά ε, θρησκευτική ελευθερία χωρίς να αφήνουμε στους πιστούς τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις απόψεις τους στους άλλους με έναν τρόπο που πραγματικά τους πείθουν και τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν την ίδια πίστη. Η απάντηση δεν είναι στον αποκλεισμό των εκφραστικών μέσων, στην ε, θύμωση της έκφρασης ε, δημοσία, αλλά να υπάρχει μια ισοτιμία στην έκφραση ε, μεταξύ αυτών που θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους και μεταξύ αυτών που είναι οι αποδέκτες αυτών των επιχειρημάτων. Το θέμα είναι να μην υπάρχει βέβαια η αίσθηση σε κανένα ότι πιέζεται για να συμμορφωθεί με κάποιες συγκεκριμένες θρησκευτικές πρακτικές που δεν επιθυμεί να σεβαστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε μια κουλτούρα ε, πληραλισμού, ελευθερίας ανεξιθρησκείας. Και ε, σε ό,τι αφορά αυτή την αυτορύθμιση που έλεγε ο συνομιλητής μου, το βασικό είναι ο σεβασμός. Ο σεβασμός. Ε, πολλά συστήματα θρησκευτικά ή αγνωστικιστικά πραγματικά πρεσβεύουν πράγματα που είναι αντιφατικά, ας πούμε, ε, με αυτά που λένε άλλα συστήματα. Παραδείγματος χάρη, ε, υπάρχουν άθεοι, ας πούμε, που βάζουν ε, διαφημίσεις ε, στα λεωφορεία ε, που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και οι χριστιανοί βάζουν τις αντίστοιχες διαφημίσεις που λένε ότι υπάρχει Θεός. Δεν το σχολιάζω. Το θέμα είναι ο κόσμος να εκφράζει τις απόψεις του δημοσία α, άνετα. Το θέμα είναι να υπάρχει σεβασμός της απόψεις των άλλων. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό με το να χρησιμοποιεί κανείς τις σκεφτικές πεπιθήσεις του άλλου με τρόπο προσβλητικό με χλεβαστικό τρόπο, με περιπεκτικό τρόπο, μια, ένα τέτοιο αυτοπεριορισμό ε, θα πρέπει να προαγάγει μια πλουραλιστική και ανεκτική κοινωνία προς την οποία όλοι κινούμαστε και την οποία φιλοδοξούμε να αποκτήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Εύανς. Αν ο Θεός είναι με τις δημόσιες μεταφορές, ίσως μπορεί να σώσουμε τον πλανήτη. Ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση για την ελευθερία έκφρασης και θρησκευτική ελευθερίας. Θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Στα πλαίσια της ε, ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης, της μεσογειακής, ευρωμεσογειακής κοινοβουλευτικής συνέλευσης, και επειδή θα συζητηθεί και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα επανέλθουμε ούτω ή άλλως. Τώρα πάμε στο σημείο 5. Έφτασαν εδώ οι εκπρόσωποι της υποομάδας για την διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Καμπότζη. Η Καμπότζη είναι μια χώρα την οποία συζητήσαμε πολλές φορές. Έχουμε υιοθετήσει ψηφίσματα που καταδίκαζαν την καταπίεση των εργαζομένων, των δημοσιογράφων, των ε, εκπροσωπών των ε, συνδικάτων και των ε, εθνικών μειονοτήτων. Πρόσφατα, μάλιστα, η τελευταία μας ακρόαση έγινε στις 23 Αυγούστου. Πολύ ωραία. Σήμερα, στα πλαίσια των συμφωνιών εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καμπότζης, υπάρχουν διάφορα εργαλεία και συζητήσεις εν εξελίξη η αντιπροσωπεία που έρχεται εδώ από την υποομάδα ε, διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα έρχεται εδώ για να, σε μια ημερίδα μελέτης ε, κατόπιν προσκλήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαιρόμαστε που θα της δώσουμε τον λόγο, αλλά ίσως καταρχήν η Γενική Διεύθυνση Ρελέξ θα μας παρουσιάσει ε, το πρόγραμμα αυτό μελέτης. Η κυρία Ντανιέλ Νταλμολάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που δεχόσαστε την ομάδα αυτή. Στη συνεδρίαση του Αυγούστου είχα μιλήσει γι' αυτό. Στα πλαίσια της συμφωνίας έχω μία ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είχαμε συμφωνήσει ότι θα ήταν ε, σημαντικό να συνεχίσουμε το διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών και να γίνει και μία διάσκεψη. Η διάσκεψη έγινε στην Καμπότζη το Νοέμβριο με μεγάλη επιτυχία, με 30 περίπου εκπροσώπου από την κυβέρνηση που συμμετείχαν σε ένα ανοιχτό και επικοδομητικό διάλογο για θέματα αφήσιμα με την κοινωνία των πολιτών. Εμείς προσκαλέσαμε αυτούς, αυτά τα άτομα να έρθουν εδώ στην Ευρώπη για να γίνει και εδώ αυτός ο διάλογος, για να μας πούν ποιες είναι οι διεκδικήσεις τους, τι προβλήματα έχουν, γιατί αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα θέλαμε να θέσουμε με την κυβέρνηση, να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση και με οικονομικά μέσα. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα που συνδέονται με, την, τα ανθρώπινα δικαιώματα, προβλήματα διακυβέρνηση, προβλήματα της συμμετοχής ε, τη κοινωνία των πολιτών στη διακυβέρνηση και στην αποκέντρωση της χώρας, προβλήματα που τέθηκαν και στις τελευταίες εκλογές, εξάλλου το είδαμε αυτό, συνεχίζεται ο εκδημοκρατισμός της χώρας, αλλά συνεχίζεται με αργό τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμετείχε ως παρατηρητής στις εκλογές του Ιουλίου και έκανε και κάποιες συστάσεις. Αυτές οι συστάσεις αποτελούν ένα τμήμα του σχεδίου δράσης στις σχέσεις μας με την καμποτζιανή κυβέρνηση αλλά και με την ε, κοινωνία των πολιτών της Καμπότζης. Από το 2003 έχουμε συγχρηματοδοτήσει διάφορα προγράμματα που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, έχουμε δώσει 9,3 εκατομμύρια και θα συνεχίσουμε με τα θέματα που μας ανησυχούν, κυρίως το θέμα της ε, ελευθερίας έκφρασης των δημοσιογράφων και των ρεπόρτερ, των ανθρώπων του τύπου εν γέννη, το πρόβλημα των εξώσεων των ιδιοκτητών, ιδιωτών και διάφορα άλλα θέματα. Δεν θέλω να σας τα αναφέρω όλα εδώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μας δώσετε αυτή την ευκαιρία. Καλό θα ήταν να αφήσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της υπόμαδα να μας πούν ποιε είναι οι ανησυχίε και τα προβλήματά τους. Ευχαριστώ και εγώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρσίντα που δουλεύει στην Κομισιόν για τον πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση και τον κοινωνία των πολιτών. Um, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα λόγια που κατά βάση το σεμινάριο του Νοεμβρίου στην Πνομπένχ και θα σας αναφέρω κάποια χοντρικά συμπεράσματα. Έχω κάνει και μια σύνοψη των βασικών σημείων ως μια χώρα η οποία από το το 1 τέταρτο του πληθυσμού της να δολοφονείται. Η Καμπότζη έχει τεράστιες λήψεις. Ως μια τραυματισμένη κοινωνία που έχει περάσει πολύ μεγάλες καταστροφές και αναταραχές, έχει δει την ε, καταστροφή των ε, νομικών και πολιτικών της ε, θεσμών. Στιγματίζεται από ανομία, δεν ισχύουν πλέον οι συνθισμένοι κανόνες συμπεριφοράς, η διαφορά ανθεί. Τα τελευταία χρόνια όμως ε, είχε κάποια επιτεύγματα. το 1993 γίνονται τακτικές εκλογές και η βία συνεχώς μειώνεται. Έχει πρώτες ύλες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξυλία και μέταλλα. Η οικονομία έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά βεβαίως υπάρχει ανησυχία πως εάν δεν αναπτυχθεί σωστά το νομικό πλαίσιο, ο πληθυσμός δεν θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί αυτές τις ε, φυσικές πηγές ήδη ακούγονται φήμες για αρπαγή γης και δωροδοκία επισήμων όσον αφορά την εκμετάλλευση αυτών των φυσικών πόρων. Το σεμινάριο μας αφορούσε τρεις βασικούς ε, Το ένα αφορούσε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, δεύτερον ο νόμο κατά διαφθοράς και τρίτον δημοκρατία και διαδικασία εκλογική, ειδικά σε σχέση με την αποστολή παρατήρησης των εκλογών. Βεβαίω αν και το κράτος της Καμπότζης ε, έχει αναγγείλει από το 1995 πως θα περάσει ένας νόμος ε, περί μη κυβερνητικών οργανώσεων, δεν υπάρχει πρόοδος. Φαίνεται πως ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τις υπηρεσίες δεν έχουν πρόβλημα, αλλά όσοι ε, σαρασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα παρενοχλούνται συστηματικά. Η τωρινή κυβέρνηση που ανέλαβε τη θητεία της τον Ιούλιο του 2008 επανέλαβε την θέλησή της να περάσει τέτοιο νόμο ο οποίο θα αποτελούσε βεβαίω ένα εργαλείο στον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Θα υπήρχε ένα μέτρο λόγοδοσίας και αυτορύθμισης, κάτι το οποίο συζητείται ήδη από τις ομάδες ε, της κοινωνίας των πολιτών και διάφορες οργανώσεις συλλογικές. Ο νόμος καταπολέμησης της ε, διαφθοράς προτάθηκε το 1994, αναδιατυπώθηκε το 2006, αλλά δεν έχει έρθει στην Εθνοσυνέλευση για έγκριση. Αναμένει την έγκριση του ποινικού κώδικα και του προϋπολογισμού. Όλοι είχαν συμφωνήσει πως ήταν απαραίτητος αυτός ο νόμος για να καταπολεμηθεί η διαφθορά στην Καμπότζη, που επίσης θα έπρεπε να ακολουθεί από μια στρατηγική εκπαίδευσης, πρόληψης και επιβολής του νόμου. Επίσης υπήρχε συμφωνία μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών πως το νομοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα των συγκρόμενων συμφερόντων, να υπάρχει προστασία των μαρτύρων και βεβαίως η δυνατότητα να υπάρξει ένα πόθεν έσχες. Φαίνεται λοιπόν πως οι απόψεις συγκλίνουν εντός και εκτός κυβέρνησης για κάτι τέτοιο. Βεβαίω αυτό θα γινόταν μέσω του να υπάρχει μια ανεξαρτησία όσον αφορά τα οικονομικά μέσα για να μην είναι οι ε, οργανισμοί αυτοί ευάλωτοι. Βεβαίως ε, ένας τρόπος θα ήταν να υπάρχει ένα εφάπαξ ετήσιο ποσό που θα δίνονταν σε αυτό τον φορέα καταπολέμησης της ε, διαφθοράς. Βεβαίως η άποψη της κυβέρνησης ήταν η απόβαση να ληφθεί από την Εθνοσυνέλευση. Βεβαίως η κοινωνία των πολιτών θέλει να προστατεύσει τις ε, πρώτε ύλε από την διαφθορά και την διαφθαρμένη εκμεταλλευσή του που στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε εκτοπισμό ανθρώπων και στην ε, εξαγωγή και την εκμετάλλευση ορυκτών μεταλλευμάτων χωρίς κανένα όφελος για τον τοπικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα, τα ευρήματα των παρατηρητών των εκλογών του 2008 και οι εξελίξει των τελευταίων ετών έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για την πρόοδο της Καμπότης προς τη δημοκρατία. Εάν ισχύσει το ίδιο για την σύσταση της επόμενης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής, καθώς ε, τα μέλη ορίζονται ανάλογα με την δύναμη των κομμάτων στην Εθνοσυνέλευση, τότε το κυβερνών κόμμα θα έχει 75% του ελέγχου αυτού του βασικού θεσμικού οργάνου. Τα μέλη της εκλογικής επιτροπής θα έπρεπε να είναι ουδέτερα, να μην ανήκουν σε κανένα ακόμα καθώς η δημοκρατική διακυβέρνηση εξαρτάται από την ύπαρξη ελέγχων και ορίων στην εξουσία. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει και απίθανο στην Καμπότζη, καθώς περνάμε προς μάλλον μια μονοκομματική κατάσταση. η σχετική συζήτηση για την εκλογική διαδικασία κατέληξε σε κάποιες ε, ανάλογες ε, συστάσεις. Όμως η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή είπε πως δια νόμου είναι ανεξάρτητη, αλλά βεβαίως στην πράξη τα πράγματα δεν είναι ποτέ τέλεια. Από την άλλη συνεργάζεται με την τεχνική αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί η διαδικασία των καταγγελιών. Οι γενικές συστάσεις λοιπόν είναι οι εξής τρεις πρώτων πρέπει να συνεχιστούν οι διάλογοι και τα σεμινάρια αυτού του τύπου το οποίο χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να αποτελέσουν τη βάση της νομικής μεταρρύθμισης. Δεύτερον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του φορέα καταπολέμησης διαφθοράς και της εκλογικής επιτροπής. Τρίτον, θα πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα για την εκλογική διαδικασία που αφορούν τους εκλογικούς καταλόγους, την πρόσβαση στα ΜΜΕ, την χρήση κρατικών πόρων και βεβαίω την βελτίωση της διαδικασίας προσφυγών. Ευχαριστώ. Okay, merci, Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η κυρία, η κυρία άρα θέλει να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω τα μέλη της αντιπροσωπείας μας στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εγώ ο ίδιος λέγομαι Τούν Σαράι, είμαι διευθυντής του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συστάθηκε το 1992. Δεύτερον, η συνάδελφος Λύση Σωτηρή, ε, διευθυντής του Κέντρου Υγείας, εκ δεξιών μου ο πρόεδρος του Εθνικού Συνδέσμου. Ε, Συγκάτ, ο γενικός ε, γραμματέας επίσης της Συγκάτ, η κυρία Ποκναντά, διευθύντρια μια μιας οργάνωσης γυναικών Διευθύντρια επίσης ε, του Κέντρου για την Μέρημνα των Παιδιών, ο κύριος Τσινχά. <laughs> Ο κύριος Πενσαμάτη, διευθυντής του, τσένος Δημοσιογράφων και επίσης της ε, διεθνής πιο δημοφιλούς ε, εφημερίδας της Καμπότζης. Ο κύριος Συντέρα, διευθυντής του Κέντρου Νομικής Εκπαίδευσης της ε, Καμπότζης. Κυρία Συντέρη, Διευθύντρια του Κέντρου Κοινωνικής Ανάπτυξης Ο κύριος Σάιουαν Σέι, διευθυντής ε, Ένωσης ε, Υποστήριξης των Μειονοτήτων. Ο κύριος Σοστέι, πρόεδρο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Νομοθεσίας. Ε, δεξιά του κύριο είναι υπεύθυνο για τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις. Ο κύριος Τσάν Σασαρότ. Ε, διευθυντής ενός προγράμματος κοινωνικής και, υποστηρι... και οικονομικής υποστήριξης. Και ο κύριος δεξιά του επίσης είναι διευθυντής ενός, μιας ένωσης νομικών. Τώρα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας παρήχε αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας αυτά τα στοιχεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού στην Καμπότζη. Ε, παλιότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποστείλει μια ομάδα παρατηρητών στις εκλογές αλλά επίσης και της περίοδου πριν και μετά τις εκλογές. Και αυτό συνέβαλε σε μια βελτίωση αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Και θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει έτσι και στο μέλλον. Ε, η κατάσταση των, κάθε φορά που η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη ε, εμφάνιζε μια επιδείνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνθηκε στην κυβέρνηση της Καμπότζη για να βελτιωθεί η κατάσταση. Θα ήθελα να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να παρατηρεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη ούτω ώστε όλοι οι πολίτε τη χώρα αυτή να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπω και οι Ευρωπαίοι πολίτε. Επίση, θα πρέπει οι πολίτε τη χώρα μα να ενταχθούν κάποια πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς στην ε, χώρα αυτή και να δοθούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα, θέλα, θα ήθελα κλείνοντας να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην εργασία σας. Bienvenue donc euh, à vous tous, euh, membres éminents euh, Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. Εάν κάποιος από εσά, από τα μέλη της αντιπροσωπείας, θα ήθελε να πάρει το λόγο για να παρουσιάσει κάποιο θέμα, παρακαλείτε να το κάνει. Bien. Est-ce que, chers euh, Ίσως ε, κάποιος από τους συναδέλφους θα ήθελε να υποβάλει κάποιες ερωτήσεις στην αντιπροσωπεία της Καμπότζη. Ο κύριο Καπάτο ίσω. Ευχαριστώ. Εγώ δυστυχώ δεν άκουσα την εισαγωγή. Θα προτιμούσα να ακούσω λοιπόν παρά να μιλήσω. Να θέσω παρόλα αυτά ένα ερώτημα και δεν ξέρω αν κανεί μπορεί να μου απαντήσει. Μάλιστα δύο ερωτήματα πιο συγκεκριμένα. Καταρχά, ποια είναι η κατάσταση των μειονοτήτων του Καμπουτσέα Κρόμ κυρίως αυτής της ε, μειονότητας. Τους γνώρισα σε μια επίσκεψη που έκανα στην Καμπότζη. Ε, ζούνε σε ιδιάλυτες συνθήκες, θα έλεγα. Ένα άλλο ερώτημα αφορά την κατάσταση των προσφύγων που φτάνουν από το Βιετνάμ. Από τις ορεινές περιοχές που φεύγουν από το Βιετνάμ και φτάνουν στην Καμπότζη. Η Καμπότζη τους επαναπατρίζει δια της βίας, ενώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα και αμφιβολίες για την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας. Επίσης υπάρχουν σοβαρότατο κίνδυνοι ε, βίας και κακομεταχείρισης όταν τα άτομα αυτά επαναπατρίζονται στο Βιετνάμ. Βέβαια αυτό αφορά και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, αλλά αφορά και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη. Γιατί δεν ξέρω αν εφαρμόζονται οι συμβάσεις του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Καμπότζη. Επίσης, ο ρόλος της ΥΠΑ της αρμοστίας ε, προσφύγων του ΟΗΕ ε, στην περιοχή είναι λίγο αμφίβολος. Α, θέλω και μια τρίτη ερώτηση. Είχα, φτάσει, πάει στην Καμπότζη στα πλαίσια μιας προεκλογικής εκστρατείας. Και πίσω από την, ε, την, τις, τις επισημότητες και τον δίθεν σεβασμό των κανόνων, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για κάθε προεκλογική εκστρατεία είναι το να γίνουν τα πράγματα, ε, να υπάρξει δηλαδή προεκλογική εξαρτία και έκφραση των κομμάτων και στην τηλεόραση. Αλλά δυστυχώς όλο τον τηλεοπτικό χρόνο τον μονοπόλησε ένα κόμμα. Επίσης υπήρξαν, παρατηρήθηκαν συλλήψει δημοσιογράφων στην προεκλογική περίοδο. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι ο έλεγχος των αρχηγών που ασκούν οι αρχηγοί των χωριών ε, σε ό,τι αφορά τις, ε, τις καταχωρήσεις στα εκλογικά μητρώα. Οι αρχηγοί των χωριών ελέγχουν πλήρως αυτές τις καταχωρήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους φιλοξενούμενούς μας μπορεί να μου απαντήσει. Τους φιλοξενούμενους αυτούς τους καλωσορίζω και εγώ. Δεν ξέρω αν κάποιος λοιπόν ε, πάνω σε αυτά τα ερωτήματα έχει κάποιες πληροφορίε να μου δώσει. Ο κ. Καπάτο είναι ο ειδικό μα για αυτά τα θέματα, βλέπετε. Ακόμα ένα ερώτημα. Η Διεθνής Αμνηστία μας μίλησε για εξώσεις ε, με στρατιωτικά μέσα, μάνου μιλιτάρι, φτωχών ανθρώπων που φεύγουν από το, την κατοικία τους χωρίς ε, αποζημίωση, χωρίς καμία πρόταση επανεγκατάστασής τους. Από ό,τι φαίνεται είναι μια πρακτική όχι καινοφανής, αν όχι συνηθισμένη, τουλάχιστον δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Υπάρχει κάποιο από εσά που γνωρίζει κάτι για την κατάσταση των ανθρώπων που έχουν ε, διωχθεί από τα σπίτια τους. I try my best to, to answer Να προσπαθήσω εγώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Η συνάδελφος εν συνεχεία θα συμπληρώσει την παρέμβασή μου για τις εξώσεις για να απαντήσω στην Πρόεδρο. Είναι ένα τεράστιο θέμα η εξώση στην κοινωνία μας. Με βάση τις πληροφορίες που έχει οργάνωσή μου, το 2008 υπήρξαν 25 περιπτώσεις αγωγών λόγω έξωσης. 10.000 ε, είναι οι οικογένειες αυτές που έχουν ε, διωχθεί ε, και 50.000 άτομα αφορούν αυτές, οι αφορούν αυτές οι πρακτικές. Η οργάνωσή μου, μάλιστα, έχει ετοιμάσει και μία έκθεση για αυτό το θέμα, στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης, ανέφερε και αυτό το θέμα και ζητά από την κυβέρνηση να σταματήσει αυτές τις πρακτικές έξωσης. Κάνουμε έκκληση επίσης στον πρέσβη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και παρόν στη συναντησή μας, και σε άλλους δωρητές από την κοινότητα των δωρητών να πιέσουν τον ε, Πρωθυπουργό μας, ούτως ώστε να μειώσει τουλάχιστον, αν όχι να σταματήσει, τουλάχιστον να μειώσει της εξώση. Και αν συνεχιστούν αυτές οι εξώσει, θα πρέπει τουλάχιστον να αποζημιώνται δίκαια αυτοί οι άνθρωποι. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Όχι μόνο το πρόβλημα της βίαιη έξωση, αλλά το πρόβλημα των αδειών για οικονομική εκμετάλλευση διαφόρων γεών. Μιλάμε για 200.000 εκτάρια σε 71 εταιρείες. Θα πρέπει, θα πρέπει επίσης να βρούμε κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους, εργατικές κατοικίες κτλ. Αλλά μέχρι στιγμής έχουν προβλεφθεί μόνο 4.000 εκτάρια. Εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την πρακτική. Μιλάμε για 10.000 οικογένειες που, θα, που επηρεάζονται από αυτή την ανάπτυξη. Μιλάμε για εταιρείε που παίρνουν από την κυβέρνηση για συμβόλαια που παίρνουν οι ιδιωτικέ εταιρείε από την κυβέρνηση. Τώρα, για του ορεσίβου αυτού που φτάνουν στην Καμπότζη. Η, Καμπότζη, η, οργάνωσή μου έχει δώσει πληροφορίε στην ύπατη αρμοστία προσφύγων. Θέλουμε να δώσουμε άσυλο σε αυτούς τους ορεσίβιου που περνάνε τα σύνορα Βιετνάμ-Καμπότζης, αλλά έχουμε κάποιες δυσκολίες, γιατί οι τοπικές οργανώσεις και εμείς που είμαστε τοπική οργάνωση αντιμετωπίζουμε εκφοβισμό από την κυβέρνηση. Εμείς δίνουμε πληροφορίες στην υπατιαρμοστία. Απλώς μόνο. Το θέμα είναι να, πάρει το, να αποκτήσει το δικαίωμα η υπατιαρμοστία να φτάσει στα σύνορα ε, και να δει αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει πληροφορίες. Ζητάμε άδεια από την κυβέρνηση για να μπορέσει η πατιαρμοστή να πάει στα σύνορα. Χρειάζεται δύο εβδομάδες συνήθως για αυτή την άδεια. Ε, σε αυτό το διάστημα όμως ε, οι τοπικές αρχές συχνά τους συλλαμβάνουν μέσα στα δάση και τους επαναπατρίζουν. Τώρα όλο και λιγότεροι άνθρωποι περνάνε τα σύνορα, γιατί υπάρχει και πίεση και προς εμάς βέβαια, αλλά και προς το Βιετνάμ ε, για το πώς ε, αντιμετωπίζουν τις μειονότητές τους. Ε, τους αναγκάζουν να ζουν μέσα σε γκέτο, Παίρνουν μάλιστα απαλωτριών τη γη του και τη δίνουν σε Βιετναμέζου. Τώρα, ό,τι ήταν να απαλωτριώσουν, τα απαλωτρίωσαν. Δεν έχουν και πολλά ακόμα να απαλωτριάσουν. Επομένω, όλο και λιγότεροι άνθρωποι περνάνε τα σύνορα προ την Καμπότζη. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο της, ε, Διεθνού, της ε, Εθνικής ε, Εκλογικής Επιτροπής. Στην προεκλογική περίοδο του 2008 προσπαθήσαμε να διορθώσουμε κάποιες από τις πρακτικές που είχαν παρατηρηθεί στις ε, δημοτικές εκλογές του 2007. Είχαν Υπήρχαν προβλήματα με τους εκλογικούς καταλόγους. Ε, περίπου 500 με 600 άνθρωποι ε, είχαν διαγραφεί από τους εκλογικούς καταλόγους, περίπου το 10%. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα με τους εκλογικούς καταλόγους. Πολλοί άνθρωποι δεν έβρισκαν το όνομά τους εκλογικούς καταλόγους το 2008 σε εκλογές και δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν λοιπόν το 2008 εξαιτία αυτού. Θα αφήσω όμως τον πρόεδρο της Εθνικής ε, Εκλογικής ε, Επιτροπής να απαντήσει στο ερώτημα για το πρόβλημα ορισμένων που δεν μπορούν να ψηφίσουν. Κυρία μου, εσείς θέλετε να προσθέσετε κάτι. Καλημέρα σε όλους. Εγώ δουλεύω με τα άστεγα παιδιά, για τα άστεγα παιδιά. Θα ήθελα να απαντήσω στο τρίτο ερώτημα. Πολύ συχνά τα παιδιά στους δρόμους πέφτουν θύματα η κυβέρνηση θέλει να καθαρίσει τους δρόμους για να είναι καθαρές οι πόλεις για τους τουρίστες. Δεν μιλάμε μόνο για τα παιδιά των μειονοτήτων. Μιλάμε για το Μπρουντίνγκ που είναι δίπλα στο Κραχάμ. Τον Ιούνιο του 2006 διάφοροι φτωχοί ε, έπεσαν θύματα των αναπτυξιακών προγραμμάτων της κυβέρνησης που τους έδιωξε από τη γη τους γιατί ήθελε να χτίσει. Καταλαβαίνετε ότι οι φτωχοί γίνονται ακόμα πιο φτωχοί. Και τα παιδιά στους δρόμους πληθαίνουν. Εγώ δουλεύω μαζί με τα παιδιά. Είμαι σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Θα ήθελα να πιέσουμε την κυβέρνηση, ούτως ώστε να σεβαστεί τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών, την οποία έχει προσυπογράψει. Γιατί όταν έχουμε προβλήματα με τις διώξεις, παράδειγμα χάρη στο Κραχάμ, τα παιδιά αυτά μένουν επί ξύλου κρεμάμενα. Εμείς καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε όλα αυτά τα παιδιά, δεν μπορούμε να τα ταΐσουμε, να τα φροντίσουμε όλα αυτά. Μπορούμε να ασχοληθούμε με ένα μικρό αριθμό παιδιών. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα παιδιά χιλιάδων οικογενειών. Στη δική μου οργάνωση ασχολούμαστε με 50 παιδιά. Τους αγοράζουμε το, σχολικό εξοπλισμό, την ποδιά τους, τα βάζουμε στα δημόσια σχολεία. Είναι δουλειά αυτή. Ε, ξοδεύουμε χρήματα. Θα ήθελα λοιπόν να φροντίσουμε τα παιδιά του δρόμου. Θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να εξακολουθήσετε να παρακολουθείτε την κατάσταση και να μας υποστηρίζετε. Αυτά, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Σοφά. Ο πρόεδρος της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Και μια και και μαζί μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, θα ήθελα να μας μιλήσει για μία από τις βασικές συστάσεις της ε, αντιπροσωπείας ε, παρατηρητών ε, στην προεκλογική περίοδο για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Παρακαλώ, ο πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε επιτρέψατε μου εξ ονόματος της Εθνικής Επιτροπής Εκλογών να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση που επέστελε αντιπροσωπεία για να, μια αντιπροσωπεία για να παρατηρήσει τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο απέστειλε κάποιους παρατηρητές, αλλά πραγματικά μας βοηθάει πολύ όσον αφορά την τεχνική συνδρομή, επί παραδείγματι, αποστέλλοντας κάποιους συμβούλους και πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα έλαβα δύο εμπειρογνώμονες για να μας βοηθήσουν στην, να βελτιώσουμε την εκλογική διαδικασία. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε ότι στις προσεχείς εκλογές θα είναι βελτιωμένη η εκλογική διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου για την ε, ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, ο κύριος Τσόγκ Σακ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ε, Τσόγκ Σακ, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Ευχαριστώ να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου. Όπως ε, ακούσατε ήδη από τον Οκτώβριο είχαμε αυτή την πιστική διαμαρτυρία και Αυτό συνέβησαν στι 25 Δεκεμβρίου 2008. Εμεί έχουμε πολλέ αποστολέ ω Δικηγορικό σύλλογο να προωθήσουμε το κράτο δικαίου, να μεταρρυθμιστεί η δημόσια διοίκηση, να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δικαιοσύνη. Και αυτή τη στιγμή στην Καμπότζη η δικαιοσύνη θα έλεγα δεν είναι 100% δίκαιη. Όπως επίσης και η διάκριση των εξουσιών στη χώρα ε, νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία. Κάποιες φορές η δικαστική εξουσία ελέγχεται από την κυβέρνηση. Οπότε ο δικηγορικός σύλλογος ζητά έντονα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει να ενισχύσουμε την δική μας ε, ε, διαχείριση πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, Να κοινού την κυβέρνηση να γίνει η νομική και δικαστική μεταρρύθμιση. Επίσης, ο δικηγορικός σύλλογος παρέχει δωρεάν νομική αρρωγή στους φτωχούς και οι δικηγόροι χωρίς σύνορα επίσης είχαν ένα ανάλογο έργο στη χώρα μας, το οποίο όμως σταμάτησε πρόσφατα και δεν έχουμε αρκετούς ε, δικηγόρους για να συνεχίσουμε αυτή τη δραστηριότητα. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Eh Ωραία λοιπόν, μετά από αυτές τις εκκλήσεις βοήθεια και τα προγράμματα αυτά που μας παρουσιάστηκαν, το λόγο έχει η Επιτροπή. Υπάρχει βούληση να γίνουν όλα αυτά, υπάρχουν τα υπόροι. Ο κύριος ε, Μορένο είμαι επιφορτισμένος με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Καμπότζη, στην Πνομπένχ και θα ήθελα πρωτίστως να σας ευχαριστήσω. Εξ ονόματος των ε, φίλων από την ε, Καμπότζη που δέχτηκαν αυτή την αντιπροσωπεία πολιτών και από την, ε, για παράδειγμα, την αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου κλπ είναι πολύ σημαντικό γιατί η Καμπότζη είναι μια χώρα ιδιαίτερα απομονωμένη και οι φίλοι αυτοί από την κοινωνία των πολιτών είχαν ίσω για πρώτη φορά την ευκαιρία να έρθουν στι Βρυξέλλε. Σήμερα το πρωί πήγαν στην Κομισιόν και θα μπορέσουν να επισκεφθούν και το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα έχουν συναντήσεις με τους εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανισμών κλπ. Εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να σπάσει αυτή η απομόνωση της χώρας αυτής που καμιά φορά έχει την εντύπωση ότι η Ευρώπη δεν ασχολείται αρκετά μαζί της. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα, θέλαμε θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έδωσε τον λόγο σε ανθρώπους όπως η κυρία αυτή που μιλάει εξ ονόματος των παιδιών ε, του δρόμου που βεβαίως αλλιώς δεν έχουν κανένα βήμα για να εισακουστεί η φωνή τους. Ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι εισακούεται η φωνή αυτών των ανθρώπων εδώ σήμερα. Δεύτερον, θα ήθελα να σα πω ότι πράγματι αυτή η αποστολή αποτελεί τμήμα ενό συνόλου δράσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή στην Καμπότζη. Και ήδη οργανώσαμε ένα σεμινάριο το οποίο αναφέρθηκε από τον εμπειρογνώμονά μας τον Νοέμβριο όπου ε, συναντήθηκαν για πρώτη φορά η Κομισιόν πόρεσε ε, να ε, οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων ε, κοινωνίας πολιτών και κυβερνητικών ε, φορέων. Χάρη σε αυτό το σεμινάριο λοιπόν ε, οι εκπρόσωποι της ε, κυβέρνησης, ακόμα και οι υφυπουργοί, μπόρεσαν να μιλήσουν με συναδέλφους που βρίσκονται και σήμερα εδώ. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό ακριβώς υπό την έννοια της προώθησης αυτής της μορφής διαλόγου. Και για ανθρώπους ειδικά που η φωνή τους δεν ακούεται είναι πολύ σημαντικό να τους δίδεται αυτή η ευκαιρία διαλόγων. Ο διάλογος αυτός είναι συνεχής γιατί δεν πρόκειται μόνο για αυτό το σεμινάριο και ή για αυτή την, τον, αυτό το γύρο επισκέψεων που κάνουν αυτή την εβδομάδα, αλλά η Κομισιόν πρόκειται να, ε, και μελλοντικά να προσπαθήσει σε σχέση με όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, δηλαδή ο νόμος κατά της διαφθοράς, ο νόμος για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ, ο νόμος σχετικά με τις αναγκαστικές εξώσεις κλπ, οι επαλατριώσεις γης, ε, όλα, για όλα αυτά τα θέματα θα προωθηθεί ο διάλογος. Τώρα, όσον αφορά τι ε, εκλογέ, αυτή η αποστολή παρακολούθηση των εκλογών πραγματικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο επειδή ήταν η πιο μεγάλη αποστολή που αριθμούσε 140 άτομα, αλλά όλη η κυβέρνηση, η κοινωνία των πολιτών, οι διεθνεί δωρητέ κλπ. Όλοι αναγνώρισαν την αξία αυτή τη αποστολή που διτύπωσε κάποιε συστάσει που αυτή τη στιγμή αποτελούν τη βίβλο, θα έλεγα, τη δική μα εργασία στη Καμπότζη και αναγνωρίζεται και από την κυβέρνηση. Οι συστάσεις λοιπόν είναι ο δικός χάρτης για την διοργάνωση των επόμενων εκλογών όπως το είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής, της Εθνικής Επιτροπής των Εκλογών, ε, είπε προηγουμένως ότι θα υπάρξει μια ομάδα Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ήδη συνήθω την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να βελτιώσουν την διοργάνωση των εκλογών που όπως ξέρετε οι εκλογές στη Καμπότζη εμφανίζουν πολλά κενά, πολλές ατέλειες. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερω είναι το πρόβλημα των τέτοιων ιδιοκτησία αυτές οι αναγκαστικές εξώσεις αυτό που συνέβη στο Κραχάμ όπου η αστυνομία και ο στρατός προέβησαν σε αυτές τις αναγκαστικές εξώσεις και σύμφωνα με τους αντιπροσώπους των ΗΠΑ στην Πνομπέν ε, αυτοί, αυτές οι αναγκαστικές εξώσεις ισοδυναμούν με κλοπή γιατί πολλούνται με, με παράνομο τρόπο αυτά τα σπίτια και δόθηκε με τον τρόπο αυτό το πράσινο φως στο Δημοτικές Αρχές Πνομπένχ να κάνει αυτές τις εξώσεις. Εγώ ως αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών δεχτήκαμε τους εκπροσώπους αυτής της κοινότητας των θυμάτων και είναι ε, κάποιοι από αυτούς παρίστανται και σήμερα εδώ και ίσως θα έπρεπε να πάρουν το λόγο για να μιλήσουν για αυτές τις αναγκαστικές εξώσεις. Και συμφωνήσαμε να ληφθούν κάποια μέτρα στο επίπεδο των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήσαμε την Προεδρία να δώσει τη συμφωνία να υπάρξει μια συνάντηση τρόικα στο επίπεδο των Υπουργών Εξωτερικών. Δεύτερον, θα υπάρξει μια επίσημη επίσκεψη των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί ακριβώς που έγιναν οι εξώσεις στα κόπεδα αυτά, στις εκτάσεις αυτές της γης όπου δεν, δεν υπάρχει ούτε πόσιμο νερό, ούτε ηλεκτρικό, ούτε τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τεράστια προβλήματα, υπάρχει το AIDS σε μεγάλα ποσοστά και είναι άνθρωποι που έχουν χάσει επίσης τη δουλειά τους 10 χιλιόμετρα μόνο από την Πνόμ Πένχα. Έτσι λοιπόν πραγματικά ασχολούμαστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το ίμιση των συναδέλφων που βρίσκονται εδώ ε, εποφελούνται από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που ε, συγχρηματοδοτούνται. Θα συνεχίσουμε αυτή την εργασία και όπως έλεγα κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής αυτής της αποστολής στην Πνομπέν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε είμαστε εδώ, θα μείνουμε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό βεβαίως που ήρθατε κι εσείς εδώ για να δείξετε την πεποίθηση ότι ο αγώνας για την ε, δρέωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να συνεχίσει. Μπράβο για την ε, θέλησή σας, τον δυναμισμό σας, τις δραστηριότητές σας. Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ. Είναι η, καλύτερη, η μεγαλύτερη επιτυχία αυτή τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε στην Καμπότζη. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. τέθηκαν κάποια ερωτήματα. Κυρίως για τις ε, μειωτικές ομάδες ε, στην Καμπότζη. Οι γηγενείς πληθυσμοί και οι μειονότητες είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οι γηγενείς πληθυσμοί είναι ε, όσοι ζουν επί αιώνες στην Καμπότζη, στα υψίπεδα και στα δάση. Οι μειονότητες είναι η Καμπουτζιοκράμ, η Κμαϊσλάμ, η τσάιντιστ. και διάφορε άλλε μειονότητες. Θα ήθελα να σα πω δύο λόγια για του γηγενεί πληθυσμού τη Καμπότζη που είναι γύρω στο 1,4 του πληθυσμού της Καμπότζης, που ήταν 14 εκατομμύρια το 1998. Αυτά είναι τα στοιχεία έχουν διαφορετικές γλώσσες, διαφορετική γλώσσα δική τους. Όλοι χρησιμοποιούν το παραδοσιακό τρόπο να δουλεύουν τη γη. Αλλά τώρα, καθώς αλλάζουν τα πράγματα, χάνουν την, τον έλεγχο στους φυσικούς πόρους που χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά εξαιτίας των απαλωτριώσεων των γεών από εξωγενείς παράγοντες, από άλλους. Επίσης υπάρχει αυτό το εθνικό σχέδιο ε, κατασκευής υποδομών στην Καμπότζη ε, και εκεί όπου μένουν οι γηγενείς πληθυσμοί. Οι αλλαγές αυτές ε, συμβαίνουν στην περιοχή των γηγενών ανθρώπων. Οι τοπικές αρχές βάζει φράγματα στους γηγενείς πληθυσμούς. Το βασικό είναι να υπάρξει αλληλεγγύη ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες, να υπάρξει προστασία της γης των γηγενών πληθυσμών. Δίδονται συμβόλαια ε, για εκμετάλλευση της γης και για εξόριξη διαφόρων στοιχείων από το έδαφος σε εθνικές και ξένες εταιρείες. Μιλάμε για γη που κανονικά ανήκε σε αυτούς τους πληθυσμούς. Έχουν δοθεί 10.000 εκτάρια μέχρι στιγμής Υπάρχει ένας νόμος ε, για την ε, γη ε, του 2001, ο οποίος εφαρμόζεται άσχημα. Υπάρχει μια δήλωση των γηγενών πληθυσμών, οι οποίοι θέλουν να, να καθυστερήσουν όλη αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία. Το Σεπτέμβριο του 2007 ε, υποστήριξαν τη σχετική δήλωση του ΟΗΕ. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους φορείς εκείνους που προστατεύουν τους γηγενείς πληθυσμούς. Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει τις ε, συμβάσει του ΟΗΕ και τις συστάσεις του ΟΗΕ για την προστασία των, της γης των ε, γηγενών πληθυσμών. Το νόμο του 2001 είχε προβλεφθεί μία διάταξη που αφορούσε την καταγραφή στο κτηματολόγιο της γης των γηγενών πληθυσμών. Αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα. Όμως οι πληθυσμοί αυτοί και η κοινωνία των, των πολιτών πιέζουν την κυβέρνηση και το αποτέλεσμα είναι ότι οι διάφοροι γηγενοί πληθυσμοί προσπαθούν να καταγραφεί η γη τους ούτως ώστε να θεωρούνται και διανόμου νόμου ιδιοκτήτες με βάση τον νόμο του 2001 Αλλά πολλοί ε, τέτοιοι πληθυσμοί δεν θεωρούν ότι ακόμη και αυτή η καταγραφή στο κτηματολόγιο δεν θα τους εξασφαλίσει τα δικαιώματά τους. Σας καταλάβαμε, λέει η Πρόεδρος. Άρα δύο λεφτά επιτρέψτε μου, λέει ο μιλητής. Οι απαλωτριώσεις αυτές γης λαμβάνουν χώρα και κυρίως απαλωτριώσεις ε, της γης των γηγενών πληθυσμών. Αυτό αφορά τη γη όλων των γηγενών πληθυσμών. Υπάρχουν απειλές, εκφοβισμοί προς τους αρχηγούς των κοινοτήτων τους. Δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις με τους πληθυσμούς αυτούς ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά προγράμματα. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει αυτές τις κοινότητες και να υποστηρίξει τον εκδημοκρατισμό στην Καμπότζη. Σας ευχαριστώ, σας καταλάβαμε. Υπάρχει η υποεπιτροπή για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γηγενών πληθυσμών. Ε, Υπάρχει και η αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ όλους. Ε, με μεγάλη χαρά σας λάβαμε εδώ και ακούσαμε τις απόψεις σας. Λοιπόν, θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της συνεδρίασής μας που αφορά ε, τα αποτελέσματα της επίσκεψης στην ε, Τουρκία της επίσκεψης αντιπροσωπείας μας στην Τουρκία. Ε, δεν ξέρω όσοι θέλουν να φύγουν και όσοι θέλουν να μείνουν, να μείνουν παρακαλώ, αλλά να μην κάνετε θόρυβο. λοιπόν, ε, ε, η παρουσίαση αυτή θα γίνει η παρουσία του κύριου Ινσέλ, ο οποίος είναι καθηγητής ε, το καθηγητής πανεπιστημίου στο Παρίσι και στο Γαλατά Σεράι στην Κωνσταντινούπολη. Je vous en prie. Ah. <laughs> on ne sait jamais avec Marco. Euh, Ωραία, λοιπόν. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Τουρκία το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, θα ζητήσουμε από τον κύριο Ινσέλκ, που είναι ανάμεσά μας σήμερα και μας έκανε αυτή την τιμή γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις στις Βρυξέλλες. Παρακαλείται λοιπόν να σχολιάσει και να μας πει ποιο είναι το παρόν επίπεδο των συζητήσεων γιατί υπήρξαν κάποιες εξελίξεις έκτοτε στην Τουρκία. Λοιπόν, θα έλεγα ότι πρώτον το γεγονός ότι πάμε κάθε χρόνο στην Τουρκία αυτό μας εξοικειώνει με ορισμένου από τους συνομιλητές μας από τη μία, από την άλλη μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε καλύτερα τις διαφορές που υπάρχουν στο, στο κλίμα και στην πολιτική συγκυρία. Ε, και τώρα θα ήθελα να πω ότι το κλίμα καθορίζεται, και ρεχείται από μια αμφιβολία στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών από τη μία και στο επίπεδο της τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά την, το πραγματικό χαρακτήρα της βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν κάπου οι διαπραγματεύσεις ένταξη της Τουρκίας. Και εγώ ως Γαλλίδα πάντοτε προσπαθώ να εξηγήσω ότι η κακοφωνία αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οφείλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπεύθυνο δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και πάντοτε σχετίζεται με την αξιοπιστία αυτή τη διαδικασίας προσχώρηση τη Τουρκία. Κατά την πρώτη επίσκεψη αντιπροσωπείας, της ε, παρανομής ε, της, ε, του ανοίγματο του πρώτου κεφαλαίου που υπήρχε ένα κλίμα δυναμικών μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Και, όπως σας είπα υπάρχει μια αμφιβολία στην Τουρκία όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών για τη βούληση των Ευρωπαίων να δεχθούν την Τουρκία. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία η οποία βαίνει αποδυναμούμενη. Ε, και για παράδειγμα ε, το σχέδιο συζήτησης για το Σύνταγμα το οποίο περιεπλάκει και υπήρχε η αίσθηση ότι η προοπτική των δημοτικών εκλογών ε, είχε αποδυναμώσει σημαντικά την βούληση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και από τη μία υπάρχει μια σωστρέφη αυξανόμενη στην Τουρκία, ένας μεγαλύτερος εθνικισμός. Και το κουρδικό πρόβλημα που είναι ένα σημαντικό νήμα στις ε, επισκέψεις μας στην Τουρκία. Το κουρδικό είναι, το εξετάζουμε σε σχέση με το πώς ε, αντιμετωπίζεται στην Τουρκία. Δηλαδή, αν ε, αντιμετωπίσετε με αυτό με όρους ασφάλειας ή της ανάγκης ενότητας του κουρδικού λαού εάν προσεγγιστεί το θέμα αυτό κάτω από αυτούς τους όρους, διατρέχει τον ε, κίνδυνο διώξεων. Αν αναπτύξει κανείς, ας πούμε, την κοινωνική, ιστορική, πολιτιστική διάσταση του κουρδικού θέματος, διατρέχει τον κίνδυνο σήμερα, ενώ κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε πριν από μία δεκαετία, διατρέχει τον κίνδυνο σήμερα, η δεν συνέβαινε με τους ίδιους όρους, ε, διατρέχει τον κίνδυνο να γίνει αντικείμενο διώξεων με το νέο άρθρο ειδικά 301 του ανανεωμένου ποινικού κώδικα που επέτρεψε σε 280 περιπτώσεις στο παρελθόν να διαφύγουν αυτό το κίνδυνο. Ε, τώρα βλέπουμε ότι η ανανέωση αυτού του κώδικα ε, δίνει δυνατότητα σε νέες διώξεις. Και βλέπουμε πολλούς εκπροσώπους του τύπου να ανησυχούν. Από τη μία γιατί ο κύριος Ερντογκάν είπε ότι δίωξε κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι αποφάνθησαν εχθρικά για το άτομό του και υπάρχουν και έντονες ε, πιέσεις άμεσες ή έμεσες μέσω φορολογικών ε, πιέσεων που επισύοντος δαμόκλια σπάθη επί του, ε, στον τύπο. Η δυνατότητα χρήσης ίντερνετ, το YouTube είναι το πιο γνωστό, έκλεισε στην Τουρκία και το θέμα αυτό επίσης διατυπώθηκε, τέθηκε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Υπουργό Εσωτερικών, το θέμα του Ιντερνετ. Ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης είναι το θέμα των βασανιστήριων. Το 2008 310 άτομα παρουσιάστηκαν στα κέντρα αποκατάσταση των θυμάτων των βασανιστήριων Ε, και ε, ήταν ε, πολλά από αυτά, 210 ήταν το 2008. Είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο λοιπόν και μια ανοιχτή υπόθεση είναι ότι ο νόμος για τις εξουσίες της αστυνομίας από τον Ιούλιο του 2007 ενθαρρύνει αυτές τις, ε, αυτούς τους οργανισμούς να, κάνουν, να προσφύγουν σε άσκηση βίας. Υπάρχουν ε, εξοδικαστικά κρούσματα βίας και αστυνομικοί, ας πούμε, ε, εφαρμόζουν την πρακτική stop and shoot. Δηλαδή λένε στα θύματα τους θα σταματήσει, θα σε πυροβολήσω. αυτή η πρακτική διευκολύνθηκε όπως σας είπα, από το νομοσχέδιο του Ιουλίου του 2007 ε, σε σχέση με τις αρμοδιότητες της αστυνομίας, τα καθήκοντα μάλλον της αστυνομίας. Επίσης, ε, ε, ψηφίκαμε μια γυναικεία φυλακή, εξαιρετικά σύγχρονη, υπερσύγχρονη στην Κωνσταντινούπολη, τόσο σύγχρονη που πραγματικά περάσαμε πάρα πολλή ώρα που να μπούμε μέσα σε αυτή την ε, φυλακή γιατί όλα είναι απολύτως αυτοματοποιημένα κλπ. Ε, χρειάστηκε λοιπόν να περάσει πάρα πολύ, ε, χρόνο για να μπούμε μέσα σε αυτή τη φυλακή. Μια φυλακή υπερσύγχρονη, υποδειγματική ά, όπου για τους όρους υποδοχή δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, μόνο ότι οι γυναίκες με τις οποίες συζητήσαμε, ή τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές, ε, δεν, δεν είχαμε να πούμε πολλά πράγματα για τις συνθήκες κράτησης, αλλά για το όσον αφορά το δικαστικό το περιεχόμενο. Δηλαδή ότι, το, το διάστημα της κράτησής τους, για παράδειγμα. Επίσης, ε, ε, Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μια πολιτική όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής των ε, μεταναστών βάσει της οποίας όσοι αλλοδαποί συλλαμβάνονται στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχοντας περάσει από την Τουρκία θα μπορούσαν βάσει αυτής της συμφωνίας η οποία ακόμα δεν υφίσταται αλλά που θα εφαρμοστεί θα μπορούσαν να αποσταλούν στην Τουρκία και να κρατηθούν εκεί σε ένα κέντρο υποδοχής αυτών των ατόμων. Και επισκεφθήκαμε λοιπόν ένα τέτοιο κέντρο και πραγματικά μας κατέπληξε οι συνθήκες που επικρατούν εκεί παρόλο που πρόκειται για ένα καινούριο κτίριο που δεν ήταν κάποιο ερείπιο παρόλα αυτά τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και η νομική βάση ε, σύμφωνα με την οποία κρατούνται αυτοί άτομα, αυτά τα άτομα ήταν εντελώς ανύπαρκτα. Δηλαδή κρατούνται πάνω από ένα χρόνο χωρίς ε, να ξέρουν σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν, για ποιο λόγο, ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει την κατάστασή τους κλπ. Ε, και τα πρόσωπα αυτά λοιπόν κρατούνται χωρίς καμία πρόσβαση σε οποιοδήποτε, ε, ούτε σε αυλή. Ε, έχουν δικαίωμα να βγουν μόνο μία ώρα ε, σε μία βλή που είναι σαν ε, πάρκινγκ. Είναι πραγματικά άθλες οι συνθήκες. Ο διευθυντής του κέντρου δεν είχε ενημερωθεί για την επίσκεψή μας, παρόλο που εμείς τον είχαμε, θελήσαμε να τον ενημερώσουμε ήταν ε, πραγματικά σαν να τον ευνηδιάσαμε ή μάλλον τον ευνηδιάσαμε και τα αποτελέσματα ήταν ολέθρια. Ε, δεν, ε, ε, όλοι ήταν στον πρώτο όροφο ήταν στιβαγμένοι οι άντρες με κρεβάτια το ένα πάνω στο άλλο και λοιπά. Δεν υπήρχε καμία αίθουσα καλά ανάγνωση σας. μην συζητάμε για κάτι τέτοιο, είναι αδιανόητο. Αλλά Ε, και όπως σας είπα πολλοί από αυτούς ε, κρατούνται πάνω από ένα χρόνο χωρίς καμία πρόσβαση στον εξωκόσμο, χωρίς κανένα δικαίωμα ε, πρόσβασης στο, στην ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες, χωρίς καμία δυνατότητα δηλαδή υποβολής αίτησης για χορήγηση ασύλου, εξαιρετικά δραματικές συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ αν περνούσα ε, μόνο δύο εβδομάδες εκεί θα τρελνόμουν. Ε, είναι σαν ένα... Το δεύτερο, ο δεύτερος όροφος ήταν σαν άσυλο. Στο τρίτο όροφο ήταν ε, οι γυναίκες. Είδαμε μια φοιτήτρια από το Μαρόκο, για παράδειγμα, την οποία είχαν μαζέψει, αυτός είναι ακριβώς ο όρος, ε, στα πλαίσια μιας επιχειρήσης Κούπα, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και που ήταν εντελώς ε, χαμένη εκεί πέρα. Ε, συζητήσαμε την κατάσταση αυτή με τον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος μας είπε ότι θα προσπαθήσει ε, να ρυθμίσει τις δυνατότητες για αυτά τα άτομα να μπορούν να συναντηθούν με τους εκπροσώπους ενός οργανισμού που να μπορεί να τους εξηγήσει τα δικαιώματά τους και να τους πει ποια είναι τα διαβήματα που έχουν να κάνουν για να βγουν από εκεί μέσα. Ε, δεσμεύτηκε λοιπόν να ρυθμίσει ο Υπουργό τουλάχιστον το θέμα αυτό και εν πάση περιπτώσει αυτό μας ε, πέτρεψε να πούμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι απολύτως παράλογο να γίνονται διαπραγματεύσεις εισδοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ υπάρχουν τέτοιου είδους κέντρα υποδοχής. Γιατί είδαμε και άλλα κέντρα χειρότερα από αυτό. Επίσης, επισκεφθήκαμε τους ομολόγους μας από την τουρκική εθνοσυνέλευση, την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Κοινοβουλίου που πραγματικά κάνουν πολύ καλή δουλειά. Ο πρόεδρός τους είναι, έχει μεγάλη θέληση, είναι ιδιαίτερος ενημερωμένος για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, κάναν, πάρα πολλές εκθέσεις και έκαναν μια έκκληση σε εμά να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις εκθέσεις αυτές στις διαπραγματεύσεις της με τον κύριο Ερντογκάν στο επίπεδο του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Εσωτερικών. Για παράδειγμα υπήρχε μια έκθεση για τη δολοφονία του Χραμ Τίνκ εκείνη την εποχή όλοι μιλούσαν σχετικά στον ε, τύπο για μια έκθεση που είχε αναθέσει ο Ερντογκάν ε, όσον αφορά την εξέταση αυτής της ε, περίπτωσης του Ντίνκ. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν είχε στα χέρια του αυτή την έκθεση. Οι έρευνες συνεχίζονταν μεν, Και υπήρχαν και άλλες ε, αντίστοιχες υποθέσεις, όχι μόνο του Ντίνκ. Euh, ο ιεραίωμένο Σαντόρο α, που είχαν σχέση με την Εργενεγκόν. Ε, ζητήσαμε λοιπόν να δημοσιευθούν αυτές οι εκθέσεις και οι έρευνες αυτές ε, να ολοκληρωθούν ούτως ώστε πραγματικά να ε, αποδιαρθωθεί το δίκτυο, αυτό το κύκλωμα αυτό, το οποίο δρά σε συνθήκες ε, ατιμορρησίας. Για να μπορέσουν να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή οι ευθύνες ε, ενδεχομένως θα βαρύνουν άτομα υψηλά ιστάμενα στο στρατό ή στο πολιτικό βίο της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν τα θέματα τα οποία θέσαμε με την ευκαιρία αυτή, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον είχαμε συναντήσει προηγούμενη, στο πλαίσιο τη προηγούμενη αντιπροσωπείας, μας φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο πρόθυμος να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Τα όσα είχε πει πριν από ένα χρόνο για, το, για την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός νέου συντάγματος κλπ. Ε, σε πολύ ψηλό επίπεδο ήταν απολύτως ε, απουσίαζε η βούληση αυτή απολύτως από τις συζητήσεις. Δεν έγινε καμία μνήα ούτε καν στο επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών πράγμα που ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν σε μερίσια διάταξη πριν από ένα χρόνο. Φαίνεται ότι κατέπεσε η προεπτική αυτή. Ε, παρόλο που εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα θεμελιώδες ε, διακύβημα, όπως είπαμε στην έντευξη τύπου που δώσαμε. Ιδού λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως ε, μπορείτε να συμπληρώσετε αν έκανα κάποια παράληψη και θα ζητήσουμε τον κύριο Ελσέν να αναφερθεί στα θέματα αυτά. Euh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, έκθεση της αντιπροσωπείας σας και νομίζω ότι σε σχέση με την ε, έκθεση της προηγούμενης χρονιάς βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία προόδου ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία αλλά υπάρχει και μία στασιμότητα, αν όχι οπισθοχώρηση σε άλλα επίπεδα. Η διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Τουρκία έτσι προχωράει, με ταλαντώσεις, μπρος πίσω. Δεν ξέρουμε γιατί μερικές φορές γίνονται κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις, ενώ κάποια άλλη χρονική στιγμή έχουμε οπισθοχώρηση. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Τουρκία για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η ύπαρξη αρχών, από τη μία, υπάρχουν οι αρχές, αλλά από την άλλη έχουμε το πρόβλημα της εφαρμογής τους που είναι εντελώς αφαίρετη. Ανάλογα με τα πρόσωπα, ανάλογα με το στάτους τους, ανάλογα με την ε, περιοχή στην οποία, από την οποία προέρχονται. Συχνά ε, άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικές περιοχές ε, υφίστανται διαφορετικές παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ενώ κάποιοι άλλοι σε άλλες περιοχές δεν έχουν πρόβλημα. Αυτό είναι, είναι μια αυθαίρετη εφαρμογή κάποιων κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ησυχία της. Πέρα από, το νόμο, από τους νόμους υπάρχει η κατάρτιση του προσωπικού, των αστυνομικών, των δικαστών, αυτών που πρέπει να εφαρμόσουν τον νόμο. Δηλαδή, πέρα από την ύπαρξη των νόμων, το θέμα είναι και η εφαρμογή του. Και εκεί που οι μεταρρυθμίσει δεν προχωράνε γοργά, είναι δυστυχώς ένας από τους τομείς είναι ο τομέας τη δικαιοσύνη. Μιλήσατε για το νέο νόμο του Ιουνίου του 2007 σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας και τις ιδιοκτικές αρχές, οι οποίοι δυστυχώς ε, επειδή δεν έχουν το επαρκές επίπεδο κατάρτισης, εφαρμόζουν αφαίρετα τον νόμο. Όλα αυτά δεν αφορούν ειδικά την Τουρκία. Απλώς ε, είναι πιο οξυμένα στην περίπτωση της Τουρκίας. Βρισκόμαστε σε μια λογική καταπολέμησης τρομοκρατίας. Αυτός ο όρος καταπολέμησης δημοκρατία δημοκρατίας ε, δικαιολογεί πάρα πολλές καθυστερήσεις, οπισθοχωρήσεις, σε αυτή τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Επίσης στην έκθεσή σας αναφέρατε τη διαβόητη έκθεση που αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά τι ευθύνες της χωροφυλακής και της αστυνομίας σε ό,τι αφορά τη μη πρόληψη της δολοφονίας, των δολοφονιών αυτών που αναφέρατε. Γιατί ξέρουμε τώρα ότι γνώριζε η αστυνομία. Τελικά δημοσιεύθηκε ατύπως όμως αυτή η έκθεση, ε, κυκλοφορεί ε, στις εφημερίδες και σε ιστοσελίδες. Η έκθεση είναι τρομακτική σε ό,τι αφορά τις ευθύνες της διοίκησης της χωροφυλακής και των υπηρεσιών πληροφοριών της αστυνομίας έδειξαν σοβαρότατη αμέλεια. Η αμέλεια που θα έλεγα ότι φτάνει μέχρι και τα επίπεδα της ενοχής. Τι είδου ενοχή δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Τουλάχιστον υπάρχει μια, σαφώς μια τεράστια αμέλεια, ένοχη αμέλεια. Διαβάζοντας αυτή την έκθεση. Γιατί ήταν Αρμένιος, το θύμα γιατί είχε προκαλέσει τη μνήμη της διοίκηση του στρατού κτλ. Δεύτερον, σε σχέση με τα όσα είπατε, τονίσατε το πρόβλημα το κουρδικό. Το πρόβλημα αυτό, το κουρδικό, είναι το κεντρικό πρόβλημα, είναι η λιδία λίθος του εκδημοκρατισμού στην Τουρκία. οι περιορισμοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επειδή υποτίθεται ότι καταπολεμούμε την τρομοκρατία, απορρέει από τη μη επίλυση του Κουρδικού. Μία μικρή πρόοδος που αναφέρεται, αλλά, αλλά υλοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου του 2009, είναι ότι οι αποστολές, ε, οι εκπομπές, συγγνώμη, στην κουρδική γλώσσα γίνονται. από το 81 μέχρι το 91 θυμηθείτε ότι τα κουρδικά δεν μπορούσε να μιλήσει κανείς στον δρόμο. Τώρα είναι πολύ σημαντικό ότι ε, μεταδίδονται εκπομπές στα κουρδικά. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τα, κουρδική γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανείς στην Τουρκία. Αυτό ανοίγει νέε προοπτικές τη αναγνώρισής της από τη διοίκηση την τουρκική κτλ. Το κουρδικό πρόβλημα είναι στριμωγμένο μεταξύ ενός δόγματος της εθνικής ενότητας. Εντάξει, καλή είναι η εθνική ενότητα, αλλά το θέμα είναι τι εννοούμε με τον όρο αυτό. Είναι ένα δόγμα, ένα έθνος, μία σημαία, ένα κράτος, μία γλώσσα. Όταν υπάρχει αυτό το δόγμα περί εθνικής ενότητας με αυτές τις τέσσερις ε, συνιστώσεις, η επίλυση του κουρδικού προφανώς είναι δύσκολη. Από την άλλη, υπάρχει ένα αίτημα έτσι, πολύ ισχυρό των Κούρδων αναγνώρισης της ύπαρξής τους, της γλώσσας τους, να μεταδίδονται οι εκπομπέ στη γλώσσα τους, να ακούγεται η γλώσσα τους κτλ. Από την άλλη, μιλήσατε για τους περιορισμούς των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές προτιμήσεις κτλ. Υπάρχει μην ξεχνάμε, ένας κοινωνικός συντριτισμός αυξανόμενος μάλιστα στην Τουρκία. Υπάρχουν επομένως ε, συμπεριφορές, ε, μη σύμμορφες, ε, σεξουαλικές, πολιτικές, ε, πολιτιστικές, ε, οι οποίες απομονώνονται, για να μην πω καταστέλλονται. Η καταστολή από τη δικαιοσύνη και την αστυνομία βασίζεται σε αυτόν τον ηθικό συντριτισμό. Ακούσαμε προηγουμένως αυτή τη συζήτηση για τη θρησκεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, το πνεύμα στο οποίο λέω όλα αυτά. Ένα άλλο στοιχείο είναι κάτι που είπατε στα συμπεράσματά σας. Είπατε ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, το 2007 και 2008 προχώρησαν δυναμικά αυτές τις χρονιές, αλλά έκτοτε υπάρχει μια υπαναχώρηση. Στην Τουρκία, στην αστυνομία, στην, ε, στην πολιτική σκηνή, στη δικαιοσύνη και στην κοινωνία των πολιτών πρέπει να γνωρίσουμε. Υπάρχουν λοιπόν ε, τάσεις υπέρ της εξοκοινοβουλευτικής άσκησης της πολιτικής εξουσίας. Με αυτό, δηλαδή, το νομικό σόφισμα η νομιμότητα που απορρέει από το Κοινοβούλιο θέλουν να την περιορίσουν. Το είδατε αυτό ό,τι αφορά την εκλογή του Προέδρου της ε, Δημοκρατίας που οδήγησε στο τελεσίγραφο του στρατού. Ο λόγος για τον οποίο οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις ε, δεν νομιμοποιούνται ε, προέρχονται από τις απόψεις αυτών των ανθρώπων που είπαν ότι ένα κανονικά εκλεγμένο κοινοβούλιο δεν έχει την νομιμότητα για να αλλάξει το Σύνταγμα ακόμη και αν έχει την πλειοψηφία. Αυτό είναι ανησυχητικό. Γιατί αυτοί που, έχουν, που λένε αυτά τα πράγματα είναι και πιο δυτικόφιλοι. Αυτό είναι ένα παράδοξο, τουρκικό παράδοξο. Οι πιο ε, Ευρωπαίοι, ας πούμε, ε, φαινομενικά είναι οι πιο αυταρχικοί. Η δίκη Εργενεγκόν είναι μια πολύ σημαντική δίκη γιατί είναι ένα τεστ για να δούμε αν η κυβέρνηση και η δικαιοσύνη θα έχουν την ε, βούληση να καθαρίσουν το κράτος από τα υπολείμματα του ψυχρού πολέμου από τη μία. Η δίκη αυτή τονίσατε πλιστάκης κυλιδώνεται από τα προβλήματα της ε, ποινική διαδικασία στην Τουρκία, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, είναι η δίκη που μπορεί να γυρίσει τη σελίδα στην Τουρκία. Η σελίδα που θα, που θα κλείσουμε θα είναι τα πραξικοπήματα. Οι δολοφονίες για κρατικούς λόγους, οι εκστρατείες πολιτικής αποσταθεροποίησης και καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει από πολύ κοντά τη διεξαγωγή αυτής της δίκης. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 301, καλά νέα. Όντως υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι σε διαδικασία δίκης. Σε ό,τι αφορά όμως τους αναφέροντες αυτής της διαβόητης αναφοράς που ζητούσε συγγνώμη στους Αρμένους, ο εισαγγελέας, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ε, την αθώωσή τους για λόγους ε, ελευθερίας έκφρασης. Δηλαδή, ο εισαγγελέας έκανε μια φιλελεύθερη ερμηνεία του άρθρου 301 που πρέπει να την τονίσουμε. Να τελειώσω με δύο παρατηρήσεις. Στην έκθεση, αν και δεν ήταν δικό σας καθήκον, υπάρχει και μια διάσταση που αφορά την εφαρμογή της θρησκευτική ελευθερίας. Όχι μόνο τον περιορισμό της θρησκευτική ελευθερίας σε ό,τι αφορά τις μη μουσουλμανικές μειονότητες, αλλά κάτι με το οποίο ασχοληθήκατε. Είναι το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία των μειονοτήτων του Ισλάμ, των Αλεβιτών, που δημιουργούν προβλήματα στην κυβέρνηση. Εκεί μπλοκάρονται τα πράγματα εκεί στην κυβέρνηση, σε επίπεδο κυβέρνησης έχουμε το μπλοκάρισμα τώρα. Επίσης, η ομίχλη που υπάρχει σε σχέση με την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας δεν διευκολύνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προαγωγή των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Υπάρχει ένα παράδοξο στην Τουρκία, ότι μέσα σε μια εκλογική προοπτική, ε, στα τέλη του Μαΐου 2009, σταματάμε τις μεταρρυθμίσεις, θα έπρεπε να είμαστε σε μια αντίθετη διαδικασία, να προχωράμε τι μεταρρυθμίσεις. Αυτή την κατάσταση τη γνωρίσαμε και το 2001, όταν η προοπτική στην ε, ένταξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ανοίξει, τότε τα, τα διάφορα πολιτικά κόμματα συναγωνίζονταν το ένα το άλλο σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν μια μικρή ευθύνη ε, σε αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στην Τουρκία για τον εκδημοκρατισμό της. Ευχαριστώ κύριε Νισελ. Ο εισαγγελία αποφάσισε να μην διώξει τους αναφέροντες. Όχι ο Υπουργό Δικαιοσύνη. Α, δεν έφτασε τον Υπουργό Δικαιοσύνη στο πράγμα. Σταμάτησε δηλαδή στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα πήρε αυτή την απόφαση να σωθώσει. Γίνεται μια συζήτηση εκτό μικροφώνου βέβαια. Και εμεί μαντεύουμε. relève de la liberté d'expression. Αποφάσισε έτσι να του αθώσει για λόγους σκεφτική ελευθερία. Τι είπε στην διάσκεψη των Προέδρων για την ανάγκη ενό νέου συντάγματο. Ε, δεν ξέρω τι περιορισμοί υπάρχουν σε επίπεδο ανώτατου δικαστηρίου. Τι είπε το ανώτατο δικαστήριο. Υπάρχουν προβλήματα με την, ε, με την εκπόνηση ενό νέου συντάγματο. Υπάρχουν τέσσερα άρθρα του συντάγματο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε απαντάει Ο Τούρκο εκπρόσωπο, ο κ. Σινσέλ, ακόμα και με την απαραίτητη πλειοψηφία. Η τάση του συνταγματικού δικαστηρίου είναι ότι τα άρθρα αυτά που δεν μπορούμε να αλλάξουμε θεωρούνται ε, ως επέκταση άλλων άρθρων. Γι' αυτό έχουμε μπλοκάρει και η ερμηνεία ορισμένων συνταγματολόγων είναι ότι για να αλλάξει ένα σύνταγμα χρειάζεται μια συνταγματική συνέλευση. Και ένα κανονικό κοινοβούλιο δεν είναι μια συνταγματική συνέλευση. Γίνεται αυτού το είδους η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σέλ. No, με συγχωρείτε που έχασα την, την συζήτηση. Έχω κάτι να προσθέσω παρά το ότι υπάρχει μετά την επίσκεψή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Με ενοχλεί η αντίδραση του Προέδρου Ερντογάν και το πόσο ανυποδέχτηκαν αφού του σηκώθηκε και έφυγε από τον Ταβός. τόσο να μην δούμε τώρα ποιος συμπεριφέρθηκε σωστά, είναι η υποδοχή που είχε στην Τουρκία. Πολύ εθνικιστική έτσι αντίδραση. Επίσης λαμβάνω email από έναν καθηγητή στην Άγκυρα ο οποίος σχολιάζει τον αντισημιτισμό στην Τουρκία δεν έχω ακούσει εγώ τίποτα σοβαρό, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έλαβα είναι πολύ εκτεταμένος ο αντισημιτισμός. Και κολλάει με τα υπόλοιπα, ξέρετε, η εβραϊκή συνωμοσία για να κυβερνήσουν ε, τη χώρα μας, ε, την Τουρκία δηλαδή εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Οπότε σχετίζεται έτσι με τον εθνικισμό προφανώς έχει τη μορφή του αντισημιτισμού. Έτσι, και μπλέκεται με την υπόθεση του Νταβός. Οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή προσπαθούν να τα μπαλώσουν εκεί διπλωματικά γιατί είναι σημαντικός παράγων στη Μέση Ανατολή η Τουρκία, θεωρείται έτσι μεσολαβητής. Αλλά οι πρόσφατες αυτές εξελίξεις είναι αποθαρρυντικές. Αυτό ήθελα να πω. Monsieur Insel, vous voulez commenter ça, le retour triomphal de oui. Monsieur Erdogan euh, Bon, la, la réaction... Ωραία λοιπόν, η αντέδραση του Πρωθυπουργού του κ. Ερντογκάν πράγματι έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό στην Τουρκία γιατί η μεγάλη πλειοψηφία της τουρκικής κοινωνίας θεωρεί ότι η πράξη του Ισραήλ στη Γάζα, ιδιαίτερος εναντί η στάση έναντι των Παλαιστινίων εν γέννη ε, αντιμετωπίζεται με μεγάλη εχθρότητα στην Τουρκία. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο αντισημιτισμός πυροδοτήθηκε από αυτή τη πράξη. Ε, πρόκειται για ένα λανθάνοντα αντισημιτισμό στην Τουρκία. Ε, το διαπιστώνουμε, μιλούμε πολύ γι' αυτό, αλλά συνήθως ο αντισηματισμός περιορίζεται στο επίπεδο, στα λόγια. Δεν υπάρχει πέρασμα στην πράξη. Ε, μεταξύ του κόσμου υπάρχει μία πλήρης ε, σύγχυσης. Ο Ερντογκάν προσπάθησε να κάνει μία διάκριση μεταξύ Εβραίων και κράτους του Ισραήλ. Ε, η έκφραση σύγχυσης είναι πολύ απλή όταν οι διαμαρτυρίες οργανώθηκαν μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, στο προξενείο του Ισραήλ, αυτό θεωρώ ότι ήταν απολύτως νόμιμο, θεμητό, αλλά όταν γίνεται διαδήλωση μπροστά σε μια συναγωγή, νομίζω ότι πραγματικά διολυσταίνει κανείς προς αυτή τη σύγχυση μεταξύ δηλαδή Εβραίων και κράτους του Ισραήλ. Και ε, υπάρχουν, υπάρχει πράγματι αυτή η διολύστηση. Ο Ερντογκάν προσπάθησε να παρθώσει αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι τέλος εμείς καταπολεμούμε το σιωνισμό που είναι μία μορφή ε, εβραϊκού εθνικισμού. Κατά δεύτερο λόγο είναι στην ακραδεξιά της Τουρκίας ήδη από τη δεκαετία του 30, από τη δεκαετία του 20 θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε αντισημιτισμός. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο, έγιναν πογκρόμ το 1934 έγιναν ε, εξώσει των θρησκευτικών ε, μειονοτήτων και των Εβραίων και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Πρόκειται για έναν αντισημιτισμό ε, τον οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε περισσότερο στην Τουρκία. Η Τουρκία ανακαλύπτει ότι δεν είναι μόνο ο αντισημιτισμός αυτός ο οποίος προκαλεί προβλήματα, αλλά κάτι πολύ πέρα από αυτό η μεγάλη πλειοψηφία της τουρκικής κοινωνίας ανακαλύπτει σήμερα ότι υπάρχει και στην Τουρκία ρατσισμός, ενώ για πολλές δεκαετίες θεωρούσαμε ότι η Τουρκία ήταν μια χώρα που δεν υπήρχε θέμα ρατσισμού. Eh Ευχαριστώ. Αύριο θα συνεδριάσει το διευρυμένο Προεδρείο, αύριο το μεσημέρι. Κλείνουμε για σήμερα. Αύριο το πρωί θα τα πούμε. Έχουμε δύο πολύ σημαντικά σημεία στη μερική διάταξη. Να είστε όλοι παρά.